νέα εκβιομηχάνηση. Σα ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η κοινή συζήτηση. Η ψηφοφορία για τι εκθέσει αυτέ θα λάβει χώρα αύριο και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Κοινή συζήτηση για την συνοχή και έχουμε διάφορε εκθέσει στα πλαίσια αυτά. Καταρχά την έκθεση τη κυρία Ταμάτου για τη βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έκθεση Βάλκαρσελ Σίσο πολιτική συνοχή και στρατηγικέ έρευνα και γενοτομία για έξυπνη εξειδικεύση. Εξαίρεση τη ε, κυρία ε, Μιχαήλοβα για την Ευρωπαϊκή Ταυτική Συνεργασία Βαλή Πρακτική και και την έκθεση τη της κυρίας Μπρέσο για τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή των Αλπαιών. Και πρώτη η Κυρία Νταμάτο, ω εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τους Σκιώδης ε, γιατί είχαμε μία καλή διαπραγμάτευση. Στην Επιτροπή Ρέτζι προσπαθήσαμε να έχουμε μία ολιστική προσέγγιση για την εφαρμογή του θέματος 3, δηλαδή της ΜΜΕ στη, στο νέο προγραμματισμό. 23 εκατομμύρια επιχειρήσεις αποτελούν το 90% όλων των επιχειρήσεων και προωθούν την καινοτομία, την απασχόληση την και δημιουργούν 100.000 θέσεις εργασίας. Στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη διαφορετικότητα των ε, ΜΜΕ. Κυρία Νταμάτο, πρέπει να επιβραδύνεται. Μιλάμε για το 93% που αφορά τις ΜΜΕ και βλέπουμε ότι γίνεται καλύτερη χρηματοδότηση 64 δις που θα γίνουν 140. Αυτό είναι πρόκριμα για να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες δυσκολίες των ΜΜΕ. Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας δυστυχώς έπνιξαν την εσωτερική ζήτηση Επίσης, το διοικητικό πλαίσιο και η γραφειοκρατία αποτελούν μια ζούγκλα όπου δεν μπορεί κανείς να προβεί σε επενδύσεις. Οι δημοπρασίες θα πρέπει να είναι διαφανής γι' αυτό ε, δεχόμαστε τη νέα οδηγία για τις νέες δημοπρατήσεις και να μην υπάρχει επιβάρυνση των ΜΜΕ. Θα πρέπει να δούμε επίσης και την καθυστέρηση πληρωμών έτσι ώστε η οδηγία να εφαρμόζεται σωστά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε οι ΜΜΕ να αποθαρρυνθούν και να μην συμμετέχουν σε προγράμματα λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στην αγορά. Κυρία Νταμάτο, σας παρακαλώ επιβραδύνετε προσπαθούν να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Σας παρακαλώ, επιβραδύνετε. Και ο κύριος Καπούτο είχε το ίδιο θέμα. Πρέπει να μεταφραστούν αυτά τα δεδομένα και καταλαβαίνετε ότι αυτό επιβραδύνει τη διαδικασία. Σας παρακαλώ να επιβραδύνετε κι εσείς. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε θα ήθελα να το λάβει υπόψη η Επιτροπή. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις μικροπιστώσεις, γιατί δυστυχώς ε, την πιστοτική ασφυξία την πλήρωσαν οι ΜΜΕ. Δυστυχώς ε, θα έχουμε να κάνουμε με μια τεράστια μαύρη τρύπα. Εάν λοιπόν υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις, δυστυχώς οι κρατικές επιδοτήσεις δεν θα, δεν θα επαρκέσουν. Θα θέλαμε λοιπόν να προωθήσουμε μια περιφερειακή πολιτική που να αφορά ειδικού τομείς όπως ε, τις ε, κατασκευές και τα ε, εφή φάσματα και εφή δίκτυα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κυκλική οικονομία που θα έχει ως στόχο τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη την πράσινη απασχόληση. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανακύκλωση και την τις κατασκευές που θα λαμβάνουν υπόψη την πράσινη και οικολογική οικονομία έχει μεγάλη σημασία να λάβουμε υπόψη το κόστος ενέργειας που είναι πολύ υψηλό για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Γι' αυτό θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τη χρήση άνθρακα. Οι ΜΜΕ θα μπορούσαν να δώσουν μεγάλες ευκαιρίες στους πρόσφυγες που θα μπουν στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να είμαστε πιο παγκοσμιοποιημένη, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον κοινωνικό ιστό των επιχειρήσεων. Σας ευχαριστούμε κυρία Νταμάτο. Και ο κύριος Σίσο έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, γνωρίζετε ότι ορισμένοι άξονες δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στην τρέχουσα θητεία έχουν σχέση με την οικονομική ανάπτυξη αφενός και με την δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης αφετέρου. Η Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία ένα εργαλείο που ονομάστηκε στρατηγικές εφηβούς εξειδίκευσης. Τι είναι αυτές οι στρατηγικές εφηβούς εξειδίκευσης. Ε, πω. Ε, αφορούν την εφαρμογή της καινοτομίας, της ε, τεχνολογικής ανάπτυξης και της έρευνας στην οικονομική πραγματικότητα και στην παραγωγική πραγματικότητα των διαφόρων ε, περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε περιοχή εντοπίζει τις αδυναμίες της αλλά και τα τούτης και με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιεί αυτές τις πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές ονομάζονται RIS ε, στηρίζονται από συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία υποχρεώνουν τα κράτη, τα, τις περιοχές, τις της Ευρωπαϊκής να καθορίσουν εκ των προτέρων τις στρατηγικές τους προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση. Αυτές οι στρατηγικές ε, ρίστρια έχουν ένα συμμετοχικό χαρακτήρα, σημαντικό συμμετοχικό χαρακτήρα, γιατί εμπλέκονται επιχειρήσεις, οι οργανώσεις των πολιτών, το κράτος βέβαια, ε, πανεπιστήμια κλπ. κλπ. Εμείς στην ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, σε μια εκθέσή μας ενθαρρύναμε την Κομισιόν να προχωρήσει, να πάει ακόμη πιο μακριά με αυτές τις στρατηγικές. Και αυτή η συγκεκριμένη έκθεση είναι το, η πρώτη που ε, αφορά αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Στη σύνταξή της ε, έλαβα υπόψη τις προτάσεις διαφόρων οργανώσεων και συλλόγων. Πολλές από αυτές εξειδικευμένες στο συγκεκριμένο τομέα. Και η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης με στήριξε και υπερψήφισε αυτή την ε, πρόταση με μεγάλη πλειοψηφία. Το αποτέλεσμα της υφοφορίας ήταν 33 ψήφοι υπέρ, 3 κατά μόνο και κατά τη διάρκεια των ε, συζητήσεων υποβλήθηκαν πολλές ε, τροπολογίες, προτάσεις κλπ. που 20 ε, συγκεκριμένα προτάσεις τροπολογίες που εμπλούτησαν την ε, έκθεση. Η έκθεση αυτή μιλά για την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις ε, προσπάθειές της προκειμένου να εξασφαλίσει ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω την ανάγκη η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία να αποτελέσουν σημαντική προτεραιότητα επενδύσεων προκειμένου το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να είναι η βάση για την στήριξη, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασία. Είναι επίσης σημαντικό να αναλυθούν οι, οι ικανότητες, οι αρμοδιότητες ε, και τα προτερήματα της κάθε περιφέρειας προκειμένου να δημιουργηθούν καινούργιες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι χρειάζεται καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις περιφερειακές αρχές μέσω προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας προκειμένου να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψεις. Τελειώνω, Πρόεδρε. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό παρατηρητήριο ε, προκειμένου να ε, θέσει στη διάθεσή μας σημαντικούς χρήσιμους δείκτες. Τέλος, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας πω ποια ήταν τα προβλήματα τα οποία εντοπίζουμε σε αυτές τις ε, στρατηγικές, όχι μόνο σε σχέση με το σχεδιασμό τους, αλλά και σε σχέση με την εφαρμογή τους. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια για τέσσερα λεπτά. Η κυρία Ισκρά Μιχαήλοβα, η συγκήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επιτροπέ, σήμερα θα σας παρουσιάσω την έκθεση η οποία συζητήθηκε και η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Περιφερειακής Πολιτικής, της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα θέματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, αυτό που ονομάζουμε πρόγραμμα Interreg. Η έκθεση περιλαμβάνει κάποια στοιχεία, τις εμπειρίες, τις καινοτομίες, τη συμβολή σε τα προγράμματα Ευρώπη 2020 και την ε, απλοποίηση των προγραμμάτων ε, περιφερειακής συνεργασίας και τις συστάσεις για το μέλλον. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η συνεργασία, η διασυνοριακή, η διεθνική συνέβαλε στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών κατά τη διάρκεια των ετών αυτών για να υπάρχουν μεταφορές γνώσης και να ενημερωθούμε καλύτερα για τα προβλήματα δικαβολογικά συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων όπως η απώλεια θέσεων απασχόλησης, εκπαίδευση κτλ. Η έκθεση επίσης αναφέρει ότι ο προπολογισμό του Ιντερεκ που είναι περίπου στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ δεν αντιπροσωπεύει παρά 2,8% του προπολογισμού της περιφερειακής πολιτικής και δυστυχώ δεν ανταποκρίνεται στις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Στην έκθεση επίσης αναφέρεται ότι το πρόγραμμα, πρόγραμμα Interreg ψηφίστηκε με αρκετή καθυστέρηση και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κινητοποιήσουν τα απαραίτητα μέσα για να πετύχουν τους στόχους τους. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση προς τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ένα σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης για να γνωρίζουμε καλύτερα τι δημιουργήθηκε στα πλαίσια, ε, είχε ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα Interreg. Επίσης θα πρέπει να δοθεί το πρόγραμμα Interreg στα πλαίσια και του σημερινού πλαισίου σε ό,τι αφορά τους μετανάστες, τον έλεγχο των ε, συνοριακών περιοχών. Στην έκθεση επίσης αναφέρεται και ο σημαντικός ρόλος και συμβόλη του Interreg και τη βελτίωση της καινοτομίας και να τονωθούν οι συνέργειες μεταξύ του ΑΡΙΕΣ e και των άλλων προγραμμάτων. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε τις δραστηριότητε μας στο θέμα της ε, έρευνας και της ανάπτυξης και να υπάρχουν και πιο πολλές συνεργείες με τον ορίζοντα 2020 και με τα ταμεία επενδύσεων. Επίσης, να αυξήσουμε τον αντίκτυπο των επενδύσεων και όλα αυτά με τη σωστή χρηματοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να αποτελέσει ένα σωστό και συνεκτικό εργαλείο πρόθεσμα. Επίσης αναφέρεται η σημασία του, της Ευρωπαϊκής Ομάδας Συνεργειών και Συνεργασίας και απευθύνει έκκληση προς τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις δυνατότητες και την αποδοτικότητα του Interreg για να κινητοποιηθούν σε διασυνοριακό επίπεδο τέτοια προγράμματα συμπεριλαμβανομένου και του νομοθετικού πλαισίου. Επίσης θα πρέπει να διαπιστώσουμε ποιε είναι οι προτεραιότητε και σε περίπτωση που είναι δυνατόν να υπάρχει και μεγαλύτερη χρηματοδότηση ιδιαίτερος για τη βελτίωση τη πολιτική συνοχή. Η έκθεση υπογραμμίζει επίση ότι υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε στα πλαίσια του Interreg για να αποτελέσουν βάση για μελλοντικά προγράμματα. Και ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει βάση της πολιτικής συνοχής του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, λέει και ο Και τέλος, τελευταία εισηγήτρια για τον πρώτο γύρο αυτό, η κυρία Μερσέντε Μπρέσο για τέσσερα λεπτά επίσης. Grazie Presidente, ε, gentile Commissaria, colleghi. Ευχαριστώ. Η πολιτική συνοχή στην οποία συζητάμε σήμερα με τους τρεις συνεισηγητές αποτελούν μία πολιτική που αφορά και τις επιχειρήσεις εκτός από τους καταναλωτές. Έχει σημασία το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με έναν από τους λίγους τομείς ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την σύνοχη αλλά και για την ε, μακροπεριοχή των Άλπαιων. Η στρατηγική ΕΟΖΑΛΠ δίνει σε αυτή τη μεγάλη περιοχή τη δυνατότητα να προβεί σε κοινέ επενδύσεις προωθώντας και μία νέα θέση και δυνατότητα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Είμαι πεπισμένη ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές θα πρέπει να συνδράμουν σε αυτή τη στρατηγική, όπως σας είπα, με την έκθεση που ψηφίσαμε οι τοπικές αρχές θα πρέπει να συνδράμουν σε αυτή την στρατηγική αν θέλουμε να φτάσουμε σε αποτελέσματα. Επίσης, σε αυτή την στρατηγική δεν θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη της περιφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά φτάσουμε σε μία προστιθέμενη αξία με βάση την προηγούμενη πείρα μας και σε κοινούς στόχους έτσι ώστε να ε, συνδράμουμε στην ανάπτυξη της περιοχής των Άλπαιων. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή έχει επιπτώσει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης 2020 θα πρέπει να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και να προωθήσουμε αυτή την στρατηγική μέσα στα πλαίσια των μακροοικονομικών σχεδίων. Αυτό θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Επίσης, η στρατηγική αυτή θα πρέπει να αποτελέσει ένα νέο μέσον για την ανάπτυξη και τις οικονομικές δυνατότητες στην περιοχή, να βοηθήσουμε στον τουρισμό, στην γαστρονομία και στην ογευσία. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να υπάρχει διάδραση των ε, μεγάλων αστικών κέντρων και των αγροτικών περιοχών καθώς και των ορεινών, έτσι ώστε να επιβιώσει αυτή η στρατηγική και να ανακάμψουν αυτές οι περιοχές. Υπάρχουν πόλοι, πόροι που δεν χρησιμοποιούνται πολύ σωστά μέχρι τούδε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία πλατφόρμα επενδύσεων για την περιοχή των Άλπαιων έτσι ώστε να συνδράμει ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μέσα στα πλαίσια της ε, πολιτικής συνοχής από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, από το ΕΦΣΙ. Έτσι θα υπάρχει συνδεσιμότητα με τον ε, υπόλοιπο κόσμο γιατί πολλές φορές υπάρχουν κενά Χρειάζονται νέες λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τον επιχειρηματικό κόσμο ο οποίος θα μπορεί να δράσει και να είναι ανταγωνιστικός. Μιλάμε για δελεαστικές περιοχές με πολλές δυνατότητες για τους νέους και στην έκθεση που ενέκρινε στην πλειοψηφία της ε, η Επιτροπή θεώρησε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ε, τοπικές υποδομές. Δεν πρόκειται για την επίλυση όλων των ε, προβλημάτων, αλλά μία δυνατότητα για την μακροπεριφέρεια αυτή. Σας ευχαριστώ και τώρα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λέγω η Επιτροπής, κύριε Κρέτου. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Χαίρομαι γιατί βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συζητητές Νταμάτο, ε, Μιχαήλοβα, Νταμάτο και Σίσο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Όπως ξέρετε ασχολούμαι με θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ για αυτές τις εξαιρετικές εκθέσεις. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη την βιώσιμη και ευφύη ανάπτυξη ιδιαίτερα για την περιοχή των Άλπαιων. Όπως γνωρίζετε, έχω στη διάθεσή μου μόνο πέντε λεπτά για να σας μιλήσω για αυτά τα θέματα. Θα προσπαθήσω να τα δω εντάχει όλα. Σε σχέση με την έκθεση Νταμάτο, σε σχέση με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, χαιρετίζουμε την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη αυτές τις ενδιάμεσες στρατηγικές για την αναθεώρηση του πλαισίου και για να υπάρχει καλύτερη απασχόληση. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ΜΜΕ με βάση τους μηχανισμούς υποστήριξης των επιμέρους επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και καινοτομία σε πολλές περιφέρειες. Συμφωνώ επίσης ότι θα πρέπει όλα αυτά τα μέσα να είναι προσβάσιμα στις ΜΜΕ. Γι' αυτό, όπως γνωρίζετε, έχω λάβει μία σειρά μέτρων για την απλούστευση του ε, πλαισίου επιχειρηματικότητας και ήδη από το Σεπτέμβριο θα εισαγάγουμε αυτό τον χρηματοδοτικό κύκλο μέσα στα πλαίσια του ecohesion για να υπάρχει καλύτερη προσβασιμότητα στην αγορά. Θα πρέπει να εξεύρουμε αυτή την ισορροπία με βάση την ανάγκη απλούστευσης και του πλήρους ελέγχου για το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Η Επιτροπή επίσης θα ζητήσει να υπάρχει μια συμμετοχική πλατφόρμα για τα σχέδια των ΜΜΕ και θα πρέπει να τονίσω ότι ήδη υπάρχει μια ειδική ιστοσελίδα στον ε, ιστότοπό μας Open Data Platform, αυτή την ονομασία φέρει, έτσι ώστε οι ΜΜΕ να έχουν μία συλλογική εικόνα για τα τεκτενόμενα σε σχέση με την έκθεση του κυρίου Σίσο για την έρευνα και την ε, καινοτομία και την ευφυή e e ανάπτυξη. Χαιρετίζω αυτή την ε, πρωτοβουλία στα πλαίσια της έξυπνης ε, εξειδίκευσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Βαλκάρθελ για αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με μεγάλες προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η στρατηγική, αυτές οι στρατηγικές έρευνας και χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση και συντονισμός των ε, προγραμμάτων και των πλατφορμών σε όλα τα επίπεδα, τα διαπεριφερειακά και διασυνοριακά καθώς και τα διεθνικά θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη αυτή την πλατφόρμα της έξυπνης εξειδίκευσης σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών ε, έρευνας. Η Ισπανία με το Ινστιτούτο της Βίλης έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προς ε, αυτό το τομέα και πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές περιφέρειες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα πλαίσια της χρηματοδότης, των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης 2020. Αφορά και το ΕΦΣΙ, αυτό το πλαίσιο και το σχέδιο Juncker. Υπ' αυτή την έννοια υπάρχει ήδη ένας οδηγός που μπορείτε να συμβουλευτείτε συμπληρωματικά. Βεβαίως δεν θα σταματήσουμε εδώ, θα συνεργαστούμε και σε άλλα επίπεδα. Θα προβούμε σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών γιατί ορισμένα κράτη-μέλη και περιφέρειες ε, έχουν περισσότερη πείρα, διαφορετική ανάπτυξη και μπορούν να διαχειριστούν ευκολότερα αυτή την, αυτά τα πλαίσια έξυπνης εξειδίκευσης. Σε σχέση με την έκθεση Μιχαήλοβα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης ε, Ρίτζιο και μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων Interreg προσπαθούμε να προωθήσουμε την διασυνοριακή εδαφική συνεργασία και έχουμε επισκεφθεί επισκεφθεί 25 χώρες. Εγώ προσωπικά έχω επισκεφθεί 25 χώρες στη θητεία μου, στη μέχρι τώρα θητεία μου των δύο ετών και πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο με ανταλλαγές πληροφοριών. Θα ήθελα να σας συγχαρώ λοιπόν για αυτή την ιδέα και συμφωνώ με τις συστάσεις σας για να φτάσουμε σε μία ε, βιώσιμη στρατηγική. Χρειάζεται αυτή η κοινή στρατηγική για να είμαστε αποτελεσματικοί σε σχέση με τα δύο αυτά μέσα, δηλαδή τις, ε, την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Φυσικά χρειάζεται και μεγάλη πολιτική δέσμευση καθώς και συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών. Δυστυχώς έχουν μπλοκάρει ορισμένα διαπεριφερειακά προγράμματα. Ελπίζω να καταφέρουμε όμως να ξανανοίξουμε μία νέα δίωδο. Επίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν περιφέρειες που χρησιμοποίησαν αυτό το κοινό πλαίσιο και γι' αυτό η υποστήριξή σας είναι ύψης της σημασίας και για εμένα προσωπικά. γιατί πολλά κράτη-μέλη ε, προσπαθούν να ορθώσουν εκ νέου εθνικά σύνορα, κάτι το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνο Σε σχέση με την έκθεση Μπρεσό για την στρατηγική για την περιοχή των Άλπαιων, θα μπορούσα να τονίσω ότι πρόκειται για μία ε, ισορροπημένη προσέγγιση του ζητήματος είχα την ευκαιρία να ε, μιλήσω για αυτή τη στρατηγική, να την προωθήσω, γιατί μιλάμε για μία από τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ, όπως ακριβώς είπατε, ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τον συντονισμό της χρηματοδότησης των χρηματοδοτικών έργων και να προωθήσουμε σχέδια σε μακροπεριφερειακό επίπεδο έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τις συναφείς συνέργειες. Όπως ξέρετε, εμείς ορίσαμε ένα νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να πληρωθούν αυτοί οι στόχοι μακροπεριφερειακή, μακροπεριφερειακή στόχη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την στρατηγική για τη Βαλτική, για την Αδριατική και άλλες ε, ενέργειες που αφορούν επιμέρους περιφέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακολουθήσει με το ρόλο της ως διαμεσολαβητή. Είμαστε εταίροι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και θα πρέπει να συνδέσουμε, τα, να υπάρχει μια συνδεσιμότητα των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, ιδιαίτερα για τις περιφέρειες που είναι λιγότερο αναπτυγμένες. και θα πρέπει η δραστηριότητά μας να οδηγήσει σε μία προστιθέμενη αξία μέσα στα πλαίσια της ενεργούς ε, επικαιροποίησης των στοιχείων και των εταιρικών σχέσεων. Ε, ζητώ συγγνώμη για τη μακρηγόρησα mm. και αναμένω τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το χρόνο για τους επόμενους ομιλητές. Τώρα περνάμε στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης. Ένα λεπτό, ο Ζερόμ Λαβριγιέ. Πρόεδρε, Επίτροπε, ευχαριστώ την Mercedes Μπρέσο για την στρατηγική για τις Άλπεις. Είναι πολύ ποιοτική η έκθεση ως ε, εισηγητής νομοθέτησης, η Επιτροπή μου που εκπροσωπώ εδώ, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, ε, εκφράζει αυτή την νομοδότησή μου. Παρότι η δική μου περιφέρεια ε, είναι μακριά από την, από την περιοχή αυτή των Άλπιων, παρόλα αυτά ξέρετε ότι δεσπόζει ο όγκος αυτός και φτάνει στο Μόνσα Μισελ. Είναι πολύ σημαντική και για την απασχόληση. Θα πρέπει η στρατηγική μας να εστιαστεί στους στρατηγικούς τομείς και γι' αυτό προτείνουμε τη δημιουργία ε, τοπικών πόλων έρευνας, ε, εμπλέκοντας και τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να εθαρρύνουμε επίσης την ε, πολυμερή ενημέρωση και την ενημέρωση για την αγορά εργασίας και την ευθυγράμμιση με την αγορά εργασίας. Θα μπορούσαν να υπάρχουν κεντρικά, ε, κέντρα ενημέρωσης και μάλιστα επιγραμμικά κέντρα ενημέρωσης. Θα μπορούσαμε να, να λάβουμε υπόψη μας διάφορες προκλήσεις, την εποχικότητα, η ελεύθερη κυκλοφορία επίση των προσώπων είναι προπόθεση για να υλοποιηθούν οι στόχοι τη οικονομική συνοχή, τη κοινωνική και εδαφική, καθώ και ε, περιβαλλοντικής περιβαλλοντική συνοχή. Επίση, να λάβουμε υπόψη μα και του ε, μετακινούμενου εργαζόμενου. Για ένα λεπτό, η κυρία Μπριάνου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα περιφερειακά θέματα είναι οριζόντια αυτή είναι η βάση της νομοδότησης της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Μην ξεχνάμε την ε, βιοπικιλότητα, τον τουρισμό, τη γεωργία, ε, τη δασοκομεία. Μην ξεχνάτε ότι η κυκλική οικονομία, οι μεταφορές, η ενέργεια, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε οριζόντια. Αυτό είναι ισχύει πολύ περισσότερο για τις ορεινές περιοχές που τις ε, παραβλέπουμε συχνά ε, προ όφελο των αστικών περιοχών. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια πλούσια περιοχή σε κουλτούρα, σε παραδόσει κτλ. Ε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στην περιοχή των Άλπων. Σήμερα λιώνουν οι πάγοι και αυτό δημιουργεί κατολιστήσεις και πλημμύρες. Είναι σημαντικό επίσης να εγκαταλείψουμε την απερίμωση γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Επίση όχι μόνο η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη ελαστικότητα και να ξεπεράσουμε λιγάκι τη γραφειοκρατική προσέγγιση για να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα των τη περιοχή αυτή. Ευχαριστώ την κυρία Μπρέσο και την ευχαριστώ επίση που έλαβε υπόψη πολλά από αυτά που θέλαμε εμεί. Ευχαριστώ. Έπρεπε να πω ότι μιλάτε εξ ονόματο τη Επιτροπή ε, Περιβάλλοντο, να με συμπαθάτε. Από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, η Δανιέλα Αγίου, για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως εισηγήτρια της νομοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών, διαφωνώ και με τη μέθοδο που υιοθετήθηκε από την κυρία Μπρέσο για την τελική γνωμοδότηση, όσο και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο που ενέκριναν οι συνυπεύθυνες ε, επιτροπές που ναι μεν τις εγκρίναμε αλλά δεν υπάρχουν στο κείμενο. Η εισηγήτρια δεν ήθελε να βάλει κανένα στοιχείο που εγκρίναμε ε, οι άλλες επιτροπές και ήθελε να κάνει τα δικά της ουσιαστικά. Νομίζω ότι δεν σέβεται έτσι τη δουλειά που κάνουν οι υπόλοιπε επιτροπές. Μην ξεχνάτε επίση ότι συμφωνούν και διάφορε πολιτικέ ομάδε με αυτά που σα λέω. Σα καλώ να λάβετε υπόψη σα τι τροπολογίε που θα ψηφιστούν αύριο λοιπόν και που περιέχουν όλα αυτά τα σημεία τα οποία προέρχονται από τα κείμενα των διαφόρων γνωμοδοτήσεων των επιτροπών που δεν ελήφθησαν υπόψη από την εισηγήτρια. Σε αυτέ τι τροπολογίε, εμεί προτείνουμε θέματα όπω την ανάγκη να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση των πολιτών σε έγγραφα που αφορούν τα έργα που χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα. τη υγεία, το περιβάλλον, που είναι θέματα προτεραιότητας, ούτω ώστε με βάση, αυτές, με βάση αυτά τα θέματα να έχουμε την πρόσβαση. Δεν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε νέα έργα που αφορούν τις ε, υποδομές μεταφορών, έω, ότου υπάρχουσες ε, υποδομές ε, δεν έχουν τύχη πλήρου εκμετάλλευσης. Επίσης, είχαμε ζητήσει να μην χρηματοδοτήσουμε υποδομέ οι οποίες επιφέρουν ε, δυσανάλογο κίνδυνο για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τους φυσικούς πόρους. Το Ρήνο Λιόν, ας πούμε. Μην ξεχνάτε αυτό το έργο, το οποίο ε, δεν το ήθελε καθόλου ο τοπικός πληθυσμός. Παρόλα αυτά, δεν του λάβατε καθόλου υπόψη στις τελικές αποφάσεις. Η Επιτροπή ε, Μεταφορών θέλαμε να προωθήσουμε τη δημόσια διαβούλευση, ούτω ώστε να σεβαστούμε τη θέληση των πολιτών και να μην δημιουργήσουμε νέα μεγάλα άχρηστα έργα τα οποία καταστρέφουν ε, και την υγεία και το περιβάλλον και προωθούν την ε, διαφθορά και ε, τι μαφιόζικε διασυνδέσει. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, εξ ονόματο τη Επιτροπή Γεωργία και Ανάπτυξη Πέθρου, για ένα λεπτό, η συνάδελφο Ουλρίκε Μιούλα. Εξέτουμε, κύριε Πρόεδρε, η Γεωργία είναι η βάση για ένα παλόμενο χώρο των Άλπαιων όπως ε, γνωρίζουμε σε πολλές χώρες και μας αρέσει. Έτσι, η γεωργία και η δασοκομεία είναι και τα θεμέλια για μια επιτυχημένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Άλπεις. Ε, μόνο αν λειτουργεί σωστά εκεί η γεωργία και η δασοκομεία θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το τοπίο, να εξασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα και να δημιουργήσουμε ε, και να διατηρήσουμε ε, την ύπεθρο για τις οικογένειες εκεί για να μην φεύγουν και να ερημώνει η ύπεθρος. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί με τη χρήση των πόρων και να προστατεύσουμε προστατεύουμε την κληρονομιά. Η στρατηγική των Άλπαιων αναγνωρίζει πραγματικά ε, την ανάγκη να απαντήσουμε στις ε, ιδιαίτερότητες περιοχής. Έτσι ενισχύουμε τον τουρισμό, ε, τη βιοτεχνία και διατηρούμε τις Άλπες και ως χώρο παραγωγής και ως χώρο οικονομίας και ως χώρο διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που κατανόησαν τα βασικά σημεία και μου επέτρεψαν στη γνωμοδότησή μου να τα συμπεριλάβω. Ευχαριστώ και έρχομαστε τώρα στους ε, ομιλητές εξ πολιτικών ομάδων από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για 1,5 λεπτό. Το λόγο έχει ο κύριο Χέτμαν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα την κυρία Μιχαήλοβα, διότι πραγματικά έδωσε μεγάλη σημασία και μας επέστησε την προσοχή στην εδαφική συνεργασία. Αυτό είναι η πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ίδια ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία είναι μια ιστορία επιτυχημένη ε, ιδιαίτερα ε, για εκείνους που συνεργάζονται διασυνοριακά. Και επίσης έχουμε και καλά έργα και βέλτιστες πρακτικές ε, στα διασυνοριακά προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά και περίτρανη απόδειξη για το πώς μπορούν να συνεργάζονται οι ε, παραμεθόριες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους, καθώς και με τρίτες χώρες. Ε, τα σύνορα έτσι κι αλλιώς είναι ένας χώρος που χρειάζονται οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να γκρεμίζουμε σύνορα και συχνά τα σύνορα προφανώ είναι στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία και προσοχή. Μετά το 2020 θα πρέπει να αποδείξουμε ότι λειτουργεί αυτή η ε, εδαφική συνεργασία και να βρει και ανταπόκριση στον προπολογισμό για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τη. Χρειαζόμαστε και μεγαλύτερη ευελιξία κατά τα άλλα στην υλοποίηση και την εκτέλεση όλων αυτών των προγραμμάτων. ιδιαίτερα περισσότερη εμπιστοσύνη χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα τη διαχείριση και τη εφαρμογή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Εξ ονόματο Σοσιαλδημοκρατών για τρία λεπτά το λόγο έχει η κυρία Ντάντσίλα. Κύριε Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι, η εδαφική συνεργασία και η πολιτική συνοχής ε, είναι η πεμπτουσία της εσωτερική αγοράς. Ε, θέλουμε να αναπτυχθεί η πεθροσκέ περιφέρεια παντού, θέλουμε να υπάρξει οικονομική ολοκλήρωση στην Ευρώπη και να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των περιφερειών μας έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα η ευρωπαϊκή αγορά. Και κάθε περιφέρεια έχει το ρόλο της να διαδραματίσει και θα πρέπει να είναι πηγή ανάπτυξης με ε, ισόρροπη κατανομή των ε, οικονομικών δραστηριοτήτων σε κάθε χώρα. Πρόσφατες αναλύσεις πραγματικά ε, έρχονται να το τεκμηριώσουν αυτό. Έχει σημασία η γεωγραφία και στην περιφερειακή πολιτική όσο πουθενά αλλού. Θα πρέπει λοιπόν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να βοηθούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση να δημιουργείται και μια δικτύωση των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Δεν υπάρχει πανάκια φυσικά για την ανάπτυξη της περιφέρειας, αλλά αν έχουμε συνεργασία, διαφάνεια, επικουρικότητα, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, τότε πραγματικά θα είμαστε σε καλό δρόμο για μια σωστή εταιρική σχέση μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Μόνο έτσι ε, θα συμμετέχει όλη η κοινωνία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο δημιουργούν 85% ε, του τζίρου ε, στην περιφέρεια. Θα πρέπει να συνεργάζονται ε, λοιπόν, τα κρατημέλη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθούνται και οι γυναίκες, οι νέες υπηρεσίες και να αυξηθεί το εισόδημα των οικογενειών δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι οι ευρωπαϊκές περιφέρειες υφίστανται την πίεση της παγκοσμιοποίησης και της κλιματικής αλλαγής. Κατά τα άλλα γυράσκει και ο πληθυσμός και πολύ περισσότερο στην Ήπεθρο και στις περιφέρειες και αυτό είναι πρόκληση. Θα πρέπει να έχουμε μια αντίστοιχη λοιπόν πολιτική συνοχή στην Ευρώπη Όλοι προσπαθούμε σε μια ενωμένη Ευρώπη να ε, δρέπουμε καρπούς ε, από την πρόοδο αυτή. Οι πόλεις μας, οι δήμοι, οι κοινότητες ε, δημιουργούν πλούτο, φέρνουν επενδύσεις στη περιφερειακή και στην τοπική πολιτική και δεν θα πρέπει εμείς να παραμείνουμε παρατηρητές όλων αυτών των προσπαθειών, πρέπει να βοηθούμε. Ευχαριστώ από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές για δύο λεπτά η κυρία Τόμασιτς. Μάλα η στρέντια από τους δέτσα, τσινε κράλεσνη της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Ναι, είναι βεβαίως η σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι σημαντική για την ανάπτυξη και για να μειωθεί η ανεργία. Δεν άκουσα ποτέ έναν πολιτικό που να είναι κατά της ανταγωνιστικότητας, αλλά ε, οι περισσότεροι το καθιστούν αυτό ανέφικτο, διότι Υπάρχουν ε, μεγάλη, ε, μεγάλος φόρτος ε, διοικητικός στην αγορά, στις επιχειρήσεις και στην αγορά και είναι ανέφικτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν όπως και το φορολογικό σύστημα που χρηματοδοτεί πολιτικές δημόσιες που είναι υπερβολικές και καμιά φορά άχρηστες. Οι ΜΜΕ θα γίνουν πιο αποτελεσματικές αν οι πολιτικοί παρεμβαίνουν λιγότερο στην εργασία τους και τους δώσουν περισσότερο περιθώριο ρυθμιστικό και μειώνοντας τον φορολογικό φόρτο και επιβάρυνση. Γι' αυτό υποστηρίζω το πρόγραμμα REFIT, το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό στην εξάλληψη των εμποδίων. Βεβαίως η εσωτερική αγορά δεν εξάλληψε αυτά τα εμπόδια, αλλά ο κανονισμός ευρωπαϊκός ήρθε να προσθεθεί ε, στους κανονισμούς τους εθνικούς που υπήρχαν. Συμφωνώ να απορροφηθούν περισσότεροι περισσότερα κονδύλια ε, κοινοτικά, αλλά ε, κυρίως ε, οι ΜΜΕ των νέων χωρών δεν έχουν τέτοια ικανότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να ανανεώσουμε, να μεταρρυθμίσουμε τους κανονισμούς ούτω ώστε τα χρήματα να διοχητεύονται σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη, διότι, μόνο, διότι τότε μόνο οι, χώρες από, οι εταιρείες από ανεπτυγμένες χώρες θα τις χρησιμοποιούν. Ευχαριστώ. Φιλελεύθερη ο κύριος Οστραβίτσιος. Αγαπητοί συνάδελφοι, για τους φιλελεύθερους οι μικρομεσές είναι πάντοτε η κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 99% όλων των επιχειρήσεων ε, και ε, δημιουργούν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασία. Νομίζω ότι τα δεδομένα αυτά είναι αρκετά για να εξηγήσουν ε, την ανάγκη απλοποίησης των κανόνων ε, την ανάγκη συνεργειών, την διαφοροποίηση πόρων για τις ΜΜΕ. Ε. Επίσης, ε, το χάσμα το πολιτιστικό ανάμεσα στις διαδικασίες των διαθροτικών ταμείων και των πρακτικών των ΜΜΕ θα πρέπει να καλυφθεί. Η πολιτική της συνοχής δεν είχε ποτέ εύκολη ζωή. Από την δημιουργία της οι κριτικές υπήρξαν συνεχείς. Ωστόσο, γνωρίζουμε όλοι ότι για την ανάπτυξη έχουν τα ταμεία αυτά τα διαρθρωτικά και επενδυτικά πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις για όλες τις χώρες. Βεβαίως ε, τα χρήματα δεν είναι η μόνη επιλογή. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλά το μέσο αυτό θα πρέπει να δράσουμε ε, για απασχόληση ε, καινοτόμο των χρησιμοποίηση των δημόσιων πόρων για προστιθέμενη αξία. Πάρα πολλά χρήματα των ταμείων συνοχής δεν χρησιμοποιούνται και τόσο πολύ για την καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους της ΓΟΕ, η Ματίνα Μίκελς, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι εκθέσεις που μας απασχολούν ε, συμπεριλαμβάνουν χωρίς καμιά αμφιβολία και ε, συνοψίζουν χρήσιμες εμπειρίες που πρέπει τώρα να μεταφραστούν στην πράξη. Αυτό σημαίνει απλούστευση, απλοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιο μικρά έργα, ε, καλύτερη συνεργασία μεγαλύτερη δυνατότητα λήψη αποφάσεων τόπου και τέλος ναι, μεγαλύτερη εγκύτητα στον πολίτη. Κάτι που θα είχε ιδιαίτερη σημασία θα ήταν να σταματήσουν οι μονομερείς και μονόπλευρες πολιτικές λιτότητες που είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη συνοχή και οποιαδήποτε επενδυτική πολιτική. Και είναι παράλογο στο κάτω-κάτω όταν παγώνουν μέσα ε, διαφορετικά και να απειλούνται χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία ότι θα τους παγώσουν τα μέσα και που έτσι και αλλιώ δεν έχουν και μεγάλο περιθώριο επενδύσεων. Τέλος, ε, οι μαζικές ε, περικοπέ ή Επιθυμίσει για περικοπές το 2017 στον προπολογισμό ιδιαίτερα της συνοχής ε, απειλούν ε, την ισότητα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά ε, το επίπεδο διαβίωσης. Καλά είναι αυτά που λέει ο Γιούνκερ για ένα καινούριο κοινωνικό πυλώνα. Ωραία ακούγονται, αλλά το μοναδικό εργαλείο που υπάρχει για να επιδεικνύει αλληλέγγυα πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η πολιτική συνοχής, δεν επιτρέπεται να περικόπτεται με τέτοιο τρόπο. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Μίχελ, και τώρα από του Πρασίνους το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Μισελ Ριβαζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση αυτή θα έπρεπε να προωθεί την ε, βιώσιμη ε, ανάπτυξη στην περιοχή των Άλπαιων και δεν έχει οικολογική φιλοδοξία στις μεταφορές και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα είμαστε αδιάλεκτοι για τα μεγάλα έργα υποδομών εάν οι τροπολογίε μα δεν γίνουν δεκτές και εμεί δεν θα ψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Ζητούμε να μην είναι πια εφικτό να υπάρξει ένα έργο υποδομών αν υπάρχει ήδη μια υποδομή που υποχρησιμοποιείται και αυτό γίνεται με το ρήνο. Και στην Γαλλία είχαμε την επιβεβαίωση από το ελεγκτικό συνέδριο ε, και από τον πρόεδρο των ε, σιδηροδρόμων ότι πρόκειται για ένα μεγάλο σφάλμα είναι η επανάληψη σε έξι φορές ακριβότερο του Περπινιό Σιντεράς. Ας για το Περπινιό Φιγκέρας, για την γραμμή αυτή κόστισε 25 εκατομμύρια για το χιλιόμετρο και για το Ρήνο. Το Ρήνο θα κοστίσει περισσότερο. Βλέπουμε ότι σήμερα η γραμμή Περπινιό Φιγκέρας έχει πτωχεύσει και βλέπουμε στην έκθεση των σιδηροδρόμων ότι οι προβλέψεις κατά 85% υπερτιμήθηκαν και των εμπορευμάτων οι φορολογούμενοι πληρώνουν τον λογαριασμό, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία και η Ισπανία κατέβαλαν 50% του προϋπολογισμού. Ζητούμε καλή διαχείριση των δημοσίων πόρων. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει αποσυμφόρηση στην περιοχή των Άλπαιων από τα βαριά φορτηγά. Θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υποδομές, τις υφιστάμενες του Σε Ευχαριστώ κυρία Ριβάλντι. Και τώρα για 1,5 λεπτό εκ μέρους της ομάδας EFTD, Καλησπέρα σας. Οι επιδοτήσεις αυτές ε, είναι ε, σπατάλη των, χρημάτων των ε, φορολογουμένων. Για να έχουμε ανάπτυξη θα πρέπει να λειτουργήσουν οι αγορές, θα πρέπει να έχουν υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικά προϊόντα. Ο ρόλος ε, των αγορών είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να δώσει και διαφάνεια. Ε, δεν είναι ιδεολόγημα αυτό που σας λέω. Όταν λειτουργούν ε, οι αγορές για το κοινό καλό, αυτό είναι πολύ ζωτική σημασία και θα πρέπει οι πολιτικοί να το προωθήσουν. Υπάρχουν πολλοί επιζήμιες κατά επιπτώσεις από τα ολιγοπόλια, τα ιδιωτικά μονοπόλια και υπάρχει νεποτισμός, ε, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή την έκθεση που φανερώνει ότι τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα η συγγήτρια. Ε, που κάτι που να είναι πραγματικός ανταγωνισμός και να μην είναι νεποτισμός, ας πούμε, και πρόθεση των φίλων. Η, το να κυριαρχεί στην αγορά δεν σημαίνει μονοπόλιο. Σημαίνει ε, ότι οι μικροί α, ε, μερικές φορές λειτουργούν ως καρτέλ. Ε, συχνά, συμβαίνει αυτό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργεί με καλές προθέσεις, αλλά δεν καταλαβαίνει φύση του προβλήματος, κατασπαταλά χρήματα και επιδεινώνει την κατάσταση. Γι' αυτό η χώρα μου καταψήφισε την, ψήφισε μάλλον για να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. για ένα λεπτό από την ομάδα ΕΝΕΦ, ο κύριος Στούγκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο μας έφερε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για τη Μολδαβία. 87 εκατομμύρια ευρώ στείλαμε και σε αυτή τη μικρή χώρα πέρσι. Μα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, Πρόεδρε. Μια χώρα που κάθε χρόνο είναι πρώτη στη διαφθορά να επιβραβεύεται με εκατομμύρια ευρώ δικά μας. Και θέλετε να συζητήσουμε για στρατηγική καινοτομία. Για να κοιτάξουμε πόσο καινοτόμα χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Δίνουμε λεφτά σε βαριά διαφθαρμένες χώρες. Κάθε χρόνο, Πρόεδρε, δεκάδες φορές βλέπουμε πώς διασπαθίζονται δημόσια κονδύλια χωρίς να τιμωρείται κανείς. Και σας ζητώ εξ των φορολογουμένων να μας πείτε πότε θα σταματήσει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, από τους μη εγγεγραμμένους τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Φουντούλης, παρακαλώ. Η αποκαλούμενη οικονομική συνοχή εντός της Ένωσης δεν είναι υπαρκτή παρά μόνο στα γραφεία και στους διαδρόμους των ευρωπαϊκών οργάνων. Αλλά ακόμα και αυτό χρειάζεται πολλή συζήτηση σημαντικότατο τομέα στον οποίο θα έπρεπε να υπάρχει στήριξη και προώθηση τη καινοτομία είναι οι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. ουσιαστικά μόνο χάρη σε αυτού του είδου τι επιχειρήσει υπάρχει το σημερινό επίπεδο διαβίωση που παρά τι τεράστιε διαφορέ από χώρα σε χώρα είναι πολύ καλύτερο από αυτό των αναπτυσσομένων χωρών. δεν μπορούμε να μιλάμε για στρατηγικέ που θα δημιουργήσουν τη βάση γνώση για βιώσιμη ανάπτυξη και υψηλή ποιότητα θέσει εργασία, όταν πολλέ από τι λάθο πολιτικέ τη Ένωση έχουν οδηγήσει σε πτώση του βιωτικού επίπεδου ειδικά στις χώρες του νότου με υποαπασχόληση και κατώτατο μισθό πείνας. μάλιστα συμφωνίες όπως η ttip θα αποτελέσουν καταστροφή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. η γενικότερη κατεύθυνση είναι λανθασμένη πάλι θα δώσετε επιχορηγήσεις με κριτήρια που μικρή σχέση έχουν με την πραγματικότητα και τις ανάγκες της αγοράς με δεδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες που σε μεγάλο βαθμό θα τις εισπράξουν οι συνήθεις ύποπτοι. εάν θέλετε πραγματικά συνοχή στις οικονομίες της ένωσης τότε απαιτείται να λάβουμε μέτρα θεσπίστε ενιαίο βασικό μισθό θεσπίστε ενιαίους φορολογικούς συντελεστές δίκαιους για όλους και καταργήστε τις επιδοτήσεις ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για την αύξηση των μισθών και για να αναπληρωθούν οι όποιες φορολογικές απώλειες. να είστε σίγουροι πως έτσι οι επιχειρήσεις θα αναπνεύσουν και θα μπορέσει να επιτευχθεί σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης. όμως για να πάρθουν τέτοια μέτρα θα έπρεπε η ένωση να ενδιαφέρεται πραγματικά για υγιείς επενδύσεις και το καλό των εργαζομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των κεφαλαιοκρατών και των πολυεθνικών. ευχαριστώ. Ακολουθούν οι υπόλοιποι τώρα. Για 1,5 λεπτό η κυρία Κλάουντια Σμιτ. Αξιότιμη κυρία Πίτροπε και κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπρέσο, την εισηγήτρια, για την αγαστή και επιτυχή συνεργασία για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Άλπαιων. Πέτυχε η έκθεση και θα ήθελα να τονίσω μερικά σημεία της αυτή τη στιγμή εδώ. Ο καθένας ο οποίος ε, διάβασε, ασχολήθηκε με αυτή την έκθεση, γνωρίζει ότι έχει επιπτώσεις σε ένα χώρο που ζουν 80 εκατομμύρια άνθρωποι σε 48 περιφέρειες και σε 7 χώρες. Όταν μια έκθεση έχει τόσο μεγάλο βεληνικέ, δεν υπάρχει χώρος για διάφορες φαντασίε των αριστερών και των πρασίνων. Προστασία του περιβάλλοντος προφανώ είναι πάρα πολύ σημαντική και κάτι στο οποίο θα πρέπει να αποσκοπούμε, αλλά δεν θα πρέπει να γίνονται όλα αυτά ερήμην των ανθρώπων. Τι να το κάνω το ωραίο αλπικό τοπίο, εάν δεν υπάρχουν άνθρωποι να ζουν εκεί, να έχουμε θέσεις εργασίας και απλώς να χαίρεται ο τουρίστας και να αναγκάζονται οι άλλοι άνθρωποι να ε, αποδημούν και να μεταναστεύουν. Είναι πολύ μεγάλο τίμημα για να συμφωνήσουμε. Άρα έχει μεγάλη σημασία να επιτρέψουμε στους ανθρώπους που ζουν εκεί να παραμείνουν στην πατρίδα τους και αυτό γίνεται μόνο με υποστήριξη και επενδύσεις. Οικονομική υποστήριξη για την οικονομία, για περισσότερες θέσεις εργασίας, για διασυνοριακό εμπόριο, ε, κυκλοφορία, διαδίκτυο ε, για μια περιοχή των Άλπαιων που να μπορέσουν να ζήσουν και να εργαστούν και επόμενες γενιές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για μισή λεπτό. Κυρία Ροντρίγκες. Eh, Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια για την έκθεση αυτή, για τη συνεργασία για την περιοχή των Άλπαιων θα πρέπει να υπάρξει κινητικότητα, μεταφορά τεχνογνωσίας, νέες εταιρικές σχέσεις. Μην ξεχνάμε τους εγγενείς κινδύνους που εμφυλοχωρούν σε αυτή την ε, περιοχή. Εγώ προέρχομαι από τη Μαδέρα. Ε, χάσαμε πάνω από 6.000 εκτάρια ε, στο Φουντσάου, στην πρωτεύουσα, λόγω των πυρκαγιών. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις χαμένες. Χάθηκαν θέσεις απασχόλησης Σκοτώθηκαν άνθρωποι σε κατολιστήσεις λόγω των κλιματικών αυτών φαινομένων. Τεράστιο ήταν το κόστος σε ευρώ λόγω το, της τραγωδίας αυτής. Πού θα κάνει κάτι η Κομισιόν για το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ την Ιταλία και την Ισπανία, τις χώρες που μας βοήθησαν, αλλά και η Κομισιόν θα πρέπει να ανασκουμποθεί Θέλουμε περισσότερο σεβασμό των περιφερειών. Υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες υστερούν, οι οποίες μειονεκτούν στην Ευρώπη και πρέπει να το λάβετε υπόψη σας. Είναι σημαντικό η Κομισιό να κάνει κάτι και να υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ούτω ώστε να βοηθηθούν αυτές οι περιφέρειες. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο συνάδελφος Σενατζότο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά παίρνω το μικρόφωνο, γιατί η έκθεση για τη στρατηγική για τις Άλπεις είναι μια προσεκτική έκθεση και ευχαριστώ την κυρία Μπρέσο για αυτήν. Λαμβάνει υπόψη δύο μεγάλα θέματα. Καταρχάς, μιλάμε για μια μακροπεριφέρεια με 80 εκατομμύρια ε, κατοίκους, τις Βόρειες Άλπεις και τις Νότιες Άλπεις, που είναι ανεπτυγμένη όχι με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την υπέροχη αλπική περιοχή που είναι χρήσιμη για όλη την Ευρώπη αλλά είναι τόσο ευπαθής, τόσο δύσκολη, ε, τόσο ανοιχτή και αντιμετωπίζει προβλήματα περίμωσης. Είναι μία περιοχή που χρειάζεται την προσοχή σας. Πρέπει να υπάρχουν ενεργές υποδομές, ε, ούτως ώστε να παράγεται πλούτος, ε, ευημερία, προσοχή στο περιβάλλον, όλα αυτά τα οποία θέλουμε. Αυτές οι ίδιες υποδομές όταν περνάνε μια τόσο ευπαθή περιοχή μπορεί να γίνουν παθητικές ε, υποδομές, ενώ σε άλλες περιοχές είναι ενεργητικές. Μην ξεχνάτε ότι είναι πολύ δύσκολη η περιοχή αυτή, είναι δύσκολο να αναπτυχθεί. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει παρόλα αυτά να εξασφαλίσουμε ένα εισόδημα σε αυτές τις περιοχές, ούτω ώστε στο μέλλον να υπάρχει πληθυσμό και όχι απερίμωση. Για να υπάρξει επιστροφή του πληθυσμού θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια στρατηγική όπως αυτή που συζητάμε σήμερα και θα εγκρίνουμε αύριο. Ικανή να βοηθήσει τους ανθρώπους και να τους δώσει το επιπλέον εισόδημα γιατί ο κόσμος φεύγει όχι γιατί δεν αγαπά τη γη του Υπάρχει αυτός ο, αυτή η αγάπη και μάλιστα έντονα. Αλλά είναι τόσο δύσκολες να ζήσει κανείς αυτές τις συνθήκες. Συχνά ακούω να γίνεται λόγος για διείσδυση εγκληματικών οργανώσεων. Το λέω έτσι με ουδέτερους ε, όρους για να μην χρησιμοποιήσω τους κλασικούς Ιταλικούς. Εμείς έχουμε τα άτομα τα οποία μπορούν να ελέγξουν την ε, τελεσφόρηση των στρατηγικών ανάπτυξης. Χρειάζεται όμως αυτή η ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό, κ. Βαν Μίλτενμπεργκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι επενδύσεις είναι βάση για την ανάπτυξη και την απασχόληση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει δισεκατομμύρια στην έρευνα και την ανάπτυξη. Γι' αυτό επενδύουμε στις ευκαιρίε για το μέλλον. Αλλά στην καινοτομία όταν επενδύει δεν σημαίνει ότι αυτόματα δημιουργούνται θέσεις εργασία. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, των ε, ιδρυμάτων, των επιστημονικών, τη κοινωνία και των κρατικών αρχών. Ακριβώ αυτό θέλουμε ε, στη στρατηγική μα για την ΕΦΗ ε, έξυπνη εξειδίκευση. Είναι θετικές οι εμπειρίες, καλά πάνε τα πράγματα, αλλά μπορούν και καλύτερα. Και δύο πράγματα. Πρώτον, οι περιφέρειες ε, διαφέρουν μεταξύ τους ε, και δεν μπορούν οι περιφέρειες να αντιγράψουν απλούστατα ε, μοντέλα ε, ανάπτυξης και success story. Χρειάζεται η κάθε περιφέρεια να βασίζεται στις ίδιες δυνάμεις, στις ίδιες ανάγκες της και τις ιδιαιτερότητές της για να απτυχθεί. Δεύτερον, η έξυπνη εξειδίκευση πραγματικά μπορεί να δέσει τεράστια όθηση σε καινοτομία, σε οικονομική ανάπτυξη στις περιφέρειες, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με τις εθνικές αρχές και να ενισχύουμε την τοπική και την περιφερική αυτοδιοίκηση, να τους δίνουμε αρκετά κονδύλια για να μπορούν να επενδύουν έτσι ε, μόνο θα κάνουμε ένα άλμα προς μια Ευρώπη πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ενάμιση λεπτό. Ο κύριος Μαλτέζε. Ξοδεύουμε 26 δισεκατομμύρια για να φτιάξουμε ένα νέο τωρίνο λιόν. Ενώ υπάρχουν ε, δίκτυα τα οποία είναι θαυμάσια και μπορούν ε, να εξυπηρετήσουν την ε, εμπορική κίνηση. Εμείς φτιάξαμε, ξοδέψαμε στην Ιταλία 6 δισεκατομμύρια για να φτιάξουμε ένα είδος φραγμάτων ε, που στην πραγματικότητα πλουτίζει τους ε, διεφθαρμένους. Θα πρέπει μην ξεχνάτε ε, ότι το Καμπανίλε είναι, μια, ένα χωριό το οποίο κατέρευσε και χρειάζονται ένα ελάχιστο, κάτι ψίχουλα για να το ξαναχτίσουμε και δεν κάνουμε τίποτα παρόλα αυτά. Κάθε χρόνο έχουμε ε, και πλημμύρες όλο και πιο καταστροφικές ε, και οι πολιτικοί οι οποίοι επισκέφτονται τόπου λένε ότι θα βοηθήσουν τις περιοχές, αλλά στην πραγματικότητα ψεύδονται. Στην πραγματικότητα αυτά τα προβλήματα θα συνεχίζονται όσο δεν σταματάμε αυτή την ανώφελη πολιτική των μεγάλων έργων. Θα πρέπει να προωθήσουμε το δημόσιο συμφέρον, κυρίως να προστατεύσουμε τη ζωή των ανθρώπων και τα, τις, ε, περιοχές αυτές, τα εδάφια αυτά. Γι' αυτό θέλω να ε, υπερψηφίσετε τις τροπολογίες ε, της έκθεσης Μπρέσο για τη χρηματοδότηση διαφανών έργων, την προστασία των ε, δημόσιων υδάτινων πόρων που θα πρέπει να παραμείνουν δημόσιοι και κατά της κατασπα... κατασπατάλησης με παράλογο τρόπο πόρων για έργα όπως το Τωρίνο Λιόν. Ευχαριστώ. Ένα μισή λεπτό, κύριε Μαραγά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνούμε με την έκθεση ε, ε, για το RIS 3, αλλά υπάρχουν μερικά σημεία που θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα δει στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Πρώτον, περισσότερη περιφέρεια, λιγότερο κράτος στη διαχείριση και στη χάραξη των προγραμμάτων. Μεγαλύτερη διάδραση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις περιφέρειες. Δεύτερον, μεγαλύτερη προσοχή στα μικρά έργα και στην πραγματική ε, ανάπτυξη των παραγωγικών ιστών των περιφερειών που περνάνε σχεδόν πάντα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τρίτον, προσοχή στον κίνδυνο το να γίνει ε, απλώς μία χήμερα για να γυρίζουν χρήματα από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό στο κρατικό κορβανά. Τέσσερα, νέα έμφαση να δοθεί στην περιφερειακή ανάπτυξη. Θα πρέπει να πρωταγωνιστούν και οι πόλεις και οι περιφέρειες και να συνδέεται το πρόγραμμα RIS3 με τις κεντρικές στρατηγικές. Μιλώ για την ενεργειακή μετάβαση, και κυκλική οικονομία, κλιματική αλλαγή. Πέντε. Εξειδίκευση δεν θα πρέπει να πει, δεν σημαίνει ότι ο καθένας εργάζεται μόνος του. Θα πρέπει οι πιο προηγμένες περιφέρειες να συνεργάζονται με τις λιγότερο προηγμένες και αυτό να κυριαρχεί. Μόνο έτσι θα αποφύγουμε να ενταθούν ακόμα περισσότερο οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Και έξι, προσοχή όταν φέρνουμε νέα χρηματοδοτικά μέσα. Αλλιώς θα γίνει και θα καταντήσει να είναι μοναδικό κριτήριο η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η κερδοφορία του προγράμματος και έτσι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες ανισορροπίες και απόκληση τελικά για σύγκληση των περιφερειών. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Φων Στόρχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα συζητούμε για την πολιτική συνοχής. Τι σημαίνει αυτό. Με επιδοτήσεις θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τις οικονομικές ανισορροπίες μεταξύ των περιφέρειων. Από το 1988 έχουν δοθεί πάνω από ένα τρεις. 350 δισεκατομμύρια ακόμα λέει μέχρι το 2020 για αναδιανομή των εκατομμυρίων και των δισεκατομμυρίων. Αυτό είναι ο τώρα στις μικρομεσαίες έρχεται να λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τους δίνουμε 140 ε, δις. Αυτή είναι η σπονδυλική στήλη, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Αυτοί παράγουν τον πλούτο που στη συνέχεια αναδιανέμουμε και τους την παίρνουμε από τη δεξιά τσέπη για να τη βάλουμε στην αριστερή θα σταματήσουμε αυτή την αναδιανομή, να σταματήσουμε την πολιτική συνοχή, να τη σταματήσουμε τώρα και να φροντίσουμε καλύτερα οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις, ακριβώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να ελαφρυθούν από άχρηστο γραφειοκρατικό ε, άχθο. Αυτό θα ήταν η υπεραξία. Η κυρία Ντονανό, ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ από την νοτιοανατολική ε, Γαλλία. Θα ήθελα να κρατήσουμε τον μεγαλύτερη δεξαμενή βιοποικιλότητα ε, που είναι η περιοχή των Άλπαιων. Εδώ και 25 χρόνια υποστηρίζω την ποιότητα ζωής των πληθυσμών και τον σεβασμό του περιβάλλοντος. Κατήγγυλα το έργο γραμμής Τύρα, Το Ρήνο. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί αυτό το έργο, Νομίζω ότι η περιοχή των Άλπαιων μπορεί να υποστηρίξει βιώσιμη ε, ανάπτυξη των δασών όπως και τη διασυνοριακή περιοχή κατά των υδρογεωλογικών και κλιματικών απειλών. Επίσης, η κτηνοτροφία, η καταπολέμηση της εξόδου από την Ήπεθρο είναι προτεραιότητος. Τούτος εχόντων των πραγμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σεβαστεί το ρόλο των τοπικών αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και την σύμβαση της περιοχής των Άλπαιων του 1991, μεταξύ των οποίων η Ελβετία έχει υπογράψει αυτήν που δεν είναι μέλος της Ένωσης. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε απέναντι στη στρατηγική της μακροένταξης που θέλει να αντικαταστήσει το εθνικό και τοπικό πλαίσιο ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Για μισή λεπτό, κύριο Τσέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η σημερινή κοινή συζήτηση αφορά τέσσερις εκθέσεις για την πολιτική συνοχή και μας ξαναδείχνει ξεκάθαρα πόσο πολυσχηδής είναι αυτή η κεντρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορεί να διαμορφώνεται όταν τα μέσα και τα μέτρα είναι στοχευμένα και προς όφελος και συμφέρον των πολιτών χρησιμοποιούνται. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην έκθεση για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Μία από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερη κυκλοφορία. Τα σύνορα πλέον δεν ε, τα αντιλαμβάνεται ο κόσμος πια τη μορφή τους, μπορούν να συνεργάζονται οι παραμεθόριες περιφέρειες μεταξύ τους, που δεν είναι και πιο προηγμένες πολλές φορές στα πλαίσια ενός κράτους μέλους. Όλα αυτά μπορεί να είναι ευεργετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα υποστηρίζει εδώ και 25 χρόνια με το πρόγραμμα Interreg. Αλλά η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία είναι κάτι παραπάνω. Υπάρχει ειδικό κανονισμός και ιδιαίτερα κονδύλια για αυτά και έχουμε και ε, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συνεργασία Συνεργασίας ένα νέο νομικό μέσο για να μπορεί να υπάρχει και θεσμικά κατοχυρωμένη συνεργασία ε, πέρα από τα ακόμα υφιστάμενα κρατικά σύνορα. Δυστυχώ ερχόμαστε να διαπιστώσουμε ότι συχνά οι πρωτεύουσε για λόγου εθνικών εγωισμών υπονομεύουν αυτή τη συνεργασία και την μπλοκάρουν σε επίπεδο διασυνοριακό. και κυριαρχεί η ένομη τάξη του κράτου μέλου που πολλέ φορέ δεν συνάδει και με εκείνη του γειτονικού τη. Άρα εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη δουλειά και ελπίζω στην την επόμενη έκθεση για τη συνοχή να μιλάμε πάλι για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και στην έκτη έκθεση συνοχή. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό ο κύριο Ντέρεκ uh, Thank you, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συζητητές και την Επιτροπή για τις συνεισφορές τους και χαιρετίζω τις εκθέσεις αυτές που συζητούμε απόψη. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνήθως οι επενδύσεις ε, συγκεντρώνονται στις υποδομές και στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε την έρευνα και την ανάπτυξη. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό θα ήταν να χρησιμοποιούνται ε, στα, τα ταμεία, τα διαρθρωτικά και τα ε, κονδύλια του ορίζον 2020 μαζί, ούτως ώστε να είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιούνται μαζί αυτά τα κονδύλια και νομίζω όλοι οι κανονισμοί μπορούν να βοηθήσουν για απλό υλοποίηση ε, και ούτω ώστε να υπάρχει μια προσέγγιση των δύο ταμείων. Θα πρέπει οι μικρομεσαίες να μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία. Όλοι υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες στις περιοχές μας. Ε, πολλοί, πολλές εποφελούνται, αλλά και πάλι πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση άλλη μια φορά νομίζω ότι οι κανονισμοί μπορούν να βοηθήσουν. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές κριτικές στις περιοχές περιφερειακές πολιτικές και ακούσαμε μερικές απόψε το βράδυ. Αλλά πολλές φορές είμαστε υπερβολικά αρνητικοί. Νομίζω ότι η περιφερειακή πολιτική είναι μια επιτυχημένη ιστορία. Έχουν δημιουργηθεί επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας και θα ήθελα καμιά φορά οι συνάδελφοι να είναι πιο θετικοί ως προς το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γκέρικε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Στη σημερινή συζήτηση για τη συνοχή συζητούμε για τη μελλοντική στρατηγική των Άλπαιων της Ένωσης. Δύο σημεία για μένα σημαντικά και θέλω να τα πω εδώ. Εξ ονόματος του κόμματος των οικογενειών το έφερα στο ECR, η δημοκρατία και η βοήθεια έτσι ώστε ο κόσμος να κάνει παιδιά. Δεν είναι μόνο οικονομία και οικολογία η Άλπης, έχει και τρίτο πυλώνα, δημογραφία, γιατί το μέλλον χρειάζεται και ανάπτυξη, αλλά χρειάζεται και παιδιά. Θα πρέπει να υπάρχει ενίσχυση, επίδομα, όποιος ε, ε θέλει να αποκτήσει οικογένεια και παιδιά χρειάζεται και βοήθεια για το τοκετό, δηλαδή μέε. Δεν υπάρχουν στις Άλπε και το βλέπουμε αυτό ότι υπάρχει πρόβλημα με τους τοκετούς ε, και ε, λείπουν μέε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Πολιτών από τον Νότιο Τυρόλο για τη βοήθεια για το τοκετό ε, και υπογραμμίζουν αυτοί, αυτό που λέμε εγώ. α ζητήσουμε από κοινού Μεε στι Άλπε. Έχουν δικαίωμα οι μητέρε μα να γεννάνε με ασφάλεια και ακόμα και Ευχαριστώ κύριε Γκέρι και τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Γιάκοφτσης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Επίτροπο για την παρουσία της, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ε, θα ήθελα να τονίσω διάφορα θέματα ενδιαφέροντα για την πολιτική συνοχή που μας απασχολούν στην κοινή συζήτηση. Για ε, να υπογραμμίσω το εξής. Η πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, κυρία Μιχαήλοβα, και η συνάδελφος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Μπρέσο, έχουν εκπονήσει εξαιρετικές εκθέσεις. Ιδιαίτερα το θέμα της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει τεράστια σημασία και τεράστιο ενδιαφέρον για μας τους φιλελευθέρους. Αλλά ακούω ότι ενδιαφέρει και τους υπολείπους αυτό το θέμα, όλες οι πολιτικές ομάδες. Γνωρίζετε ε, την περιφέρεια και τη στρατηγική για την Αδριατική και, τον, και το Ιόνιο. Ε, είναι αυτή που με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο, αλλά ας μιλήσω λίγο για τις Άλπεις. Και να σας αναφέρω ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις στρατηγικές. Εμείς Λέμε ε, για τα τρία όχι. Όχι σε νέε δομέ στι μακροπεριφέρειε, όχι στη χρηματοδότηση, όχι νέα μέσα δηλαδή. Και τρίτο όχι ε, σε νέε ε, διατάξεις και ρυθμίσεις. Υπάρχουν μακροπεριφέρειες, άρχισαν να λειτουργούν σωστά, έχουν σταθεί στα πόδια τους. Βαλτική, ε, Δούναβης, Αδριατική, Ιόνιο. Μήπως να τις αφήσουμε αυτές τις περιφέρειες να δουλέψουν και να καταργηθούν αυτά τα τρία όχι για να δουλέψουν και να επιζήσουν οι μακροπεριφέρειες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδημούλης, παρακαλώ για ένα λεπτό. Κυρία Επίτροπε, κυρία Κρέτσου, τα τελευταία χρόνια η καλησπέρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πολύ οι ανισότητες και οι κοινωνικές και οι περιφερειακές. Και αυτό απειλεί τη συνοχή της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και αυξάνει όσους δεν βλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εκπλήρωση των προσδοκιών τους. Ιδίως στις χώρες του Νότου αυτό σημαίνει ότι η πολιτική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί και όχι να αποδυναμωθεί Για τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αποδυνάμωση. Και επίσης πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια έτσι ώστε τα χρήματα από την πολιτική συνοχή και περισσότερα να γίνουν και να πάνε εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια, μεγαλύτερη ανεργία, μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες, μεγαλύτερη αποεπένδυση. Και φυσικά χρειάζεται στη χώρα μου την Ελλάδα που τις τελευταίες μέρες έχει υποστεί μια μεγάλη φυσική καταστροφή με νεκρούς, με πλημμύρες, με καταστροφές να κινηθεί επιγόντως και ταχύτερα το Ταμείο Αλληλεγγύης με βάση τους προβλεπόμενους κανονισμούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, εμείς από τη Λέγκα είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή η στρατηγική για τις Άλπεις ε, ουσιαστικά εξυπηρετεί το βορρά της Ιταλίας και τη Λομβαρδία. Νομίζω ότι είναι καθυστερημένη η απάντηση, αλλά τέλος πάντων δόθηκε και είναι σοβαρή και πολλά υποσχόμενη. Ε, από... Αυτό ο πληθυσμό των Άλπιων έχει πάρα πολλά αιτήματα. Είναι υπέροχη αυτή η περιοχή. Ε, έχει μια θαυμάσια ταυτότητα οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να δουν το χέρι της Ευρώπης, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η οποία ε, δεν έγινε πολύ αισθητή μέχρι τώρα, ε, για να δώσει και βοήθεια στη βιοπικιλότητα και ανάπτυξη. Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Διερωτώμεθα, ε, η Επίτροπος και οι συγκητές θα πρέπει να διερωτηθούν. Η πολιτική στήριξη των κρατών μελών, παραδείγματος χάρη της χώρας μας, όπου υπάρχει η κυβέρνηση Ρέντζη, που προβλέπει ε, στο Σύνταγμα να ακυρωθούν οι δυνάμεις ε, και οι αρμοδιότητες των περιφερειών. Τι πράγματα είναι αυτά. Όποιοι θα λέει αυτά θα πρέπει να ντρέπεται. Εμείς θα πρέπει να υπρασπιστούμε τις ε, αρμοδιότητες των Δήμων, κοινοτήτων, τη τοπική αυτοδιοίκηση και των περιφερειών. Για 1,5 λεπτό, Μπόγκοβιτς. Σα σας Η εισηγήτρια. Κυρία Επίτροπε, η πολιτική συνοχής έχει σαν σκοπό να μειωθούν οι διαφορές στην ανάπτυξη των περιφερειών αλλά και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον θέλει να εξασφαλίσει την ανάπτυξη και τρίτον να συνενώσει τις περιφέρειες και τα διάφορα τμήματα της Ευρώπης. Καταρχάς, θα ήθελα να μιλήσω για την έκθεση για την έξυπνη εξειδίκευση. Πρώτα απ' όλα, η Ευρώπη δεν μπορεί να εξασφαλίσει αποτελεσματική συνεργασία στην οικονομία, στην επιστήμη, στην καινοτομία και στην εξειδίκευση. Εξού και η τεχνολογική μας καθυστέρηση σε κάποια τμήματα της Ευρώπης απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν τι χρειαζόμαστε να κάνουμε. Πρέπει να επιταχύνουμε και να προωθήσουμε τα μέτρα συνοχής τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο θέμα που θέλω να αγγίξω είναι η στρατηγική για την αλπική περιοχή. Ε, είμαι Σλοβένα και είμαστε πρόεδροι της περιφέρειας των Άλπαιων του, του, του φορέα δηλαδή, που διαχειρίζεται την περιοχή των Άλπαιων, θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στου ανθρώπου που ζουν σε αυτήν την υπέροχη περιοχή να κρατήσουν αναλύωτο το τοπίο του και να κρατήσουν τη ζωή και την οικονομική δραστηριότητα μέσω τη βοήθειά μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συγγνώμη, ένα, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί ακριβώς με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πιστεύω ότι ε, θα προχωρήσουμε και έχω κάνει αντίστοιχες τροπολογίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές όπως γνωρίζουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργούν θέσεις εργασίας και μάλιστα και σε περιφέρειες απομακρυσμένες και δύσκολες και στα μικρά χωριά ακόμα. Αυτό δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, συμφωνούμε όλοι. Γι' αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες, τα κράτη-μέλη, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο που έχουν και οι μεγάλες εταιρείες. Πρόσβαση σε ε, διαγωνισμούς ε, και ίδια φορολογική μεταχείριση. Θα ήταν λοιπόν αποφασιστική σημασία για να εξυγχρονιστούν οι υπηρεσίε και να δημιουργηθούν και νέε θέσει εργασία. Επίση, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό η κείμενη νομοθεσία να εφαρμόζεται σωστά. Δεν χρειάζεται πάντα καινούργια νομοθεσία. Άρα θα πρέπει και το δημόσιο να εξοφλεί τους λογαριασμούς και τα χρέη εντός 30 ημερών, που ως γνωστόν δεν γίνεται. Δεν μπορούν οι μικρομεσαίες να υφίστανται αυτή τη γραφειοκρατία και αυτές τις καθυστερήσεις. Ε, χρειάζεται να ελαφρυνθεί αυτή η επιβάρυνση και να φύγει από όλε τι νομοθεσίε και των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ και του τέσσερι ηγητέ για τι καταπληκτικέ εκθέσει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Για ένα λεπτό, ο κύριο Όμπερ Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τη συζήτηση για τις Άλπες και την οικονομική τους ενίσχυση και ε, αναγνωρίζεται ε, η σημασία των σιδηροδρόμων και η προστασία των ιδιαίτερων πόρων. Είναι ευαίσθητη η περιοχή των Άλπαιων και θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και η προστασία της φύσης. Το λέει και η έκθεση. θα, πρέπει ε, να ενισχύουμε και την άγρια πανίδα, τους ε, λύκους, τα αρπακτικά όπως ενδιαφέρεται που είναι πολύ σημαντική για τη βιοπικιλότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρείται και το τοπίο των Άλπαιων, να το φροντίζουμε, να το ενισχύουμε και να το προφυλάσσουμε. Γι' αυτό ε, θα πρέπει ε, να σκεφτόμαστε και τους γεωργούς και τους δασοκόμους που εκείνοι εξασφαλίζουν τη ζωή στην ύπεθρο αυτή. Χρειάζονται και σωστές τιμές για τα προϊόντα τους ε, και στήριξη στη στρατηγική των Άλπων και αυτή. Ευχαριστώ κύριο Μπερμάιερ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο χώρος των Άλπαιων γενικά είναι ένα περίπλοκο σύστημα. Έχουμε σύνορα, πολιτικά σύνορα, δύσκολες διασυνδέσεις και από τουριστική σκοπιά είναι σημαντικέ οι Άλπεις αρκεί να σκεφτούμε ότι περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν διακοπές το χρόνο στις Άλπεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι το είναι ένα ε, θέρετρο αλλά και χειμερινό προορισμό στις Άλπεις υπάρχουν περιφέρειες πάρα πολύ ανεπτυγμένες και πολλές ε, φορές ε, πολύ υπανάπτυκτες περιφέρειες. Γι' αυτό είναι σωστό να έχουμε μια κοινή στρατηγική και μια κοινή στρατηγική μεταφορών και συγκοινωνιών. Και καλό είναι να φύγει από τον αυτοκινητόδρομο και να πάει στο δρόμο. Και εκεί χρειάζονται γενναίες επενδύσεις ε, και στο Μπρένερο από που κατάγομαι και στο Τωρίνο Λιόν. Γι' αυτό είμαι τελείως κατά των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Ε, ε, λοιπόν, ο χώρα, λοιπόν, χώρος μάλλον των Άλπαιων είναι ε, χώρος φύσης, χώρος πολιτισμού αλλά και χώρος οικονομίας. Από ό,τι φαίνεται θα, θέλει, θέλουν κάποιοι αναγκαστικά να φέρουν μεγάλα αρπακτικά χωρίς να μπορεί ο άνθρωπος να επεμβαίνει. Μα θα σπάσει αυτή η εύθραυστη ισορροπία και θα είναι περισσότερο υπέρ της φύσης και εις βάρος του πολιτιστικού χώρου που λέγονται Άλπης και του οικονομικού χώρου Άλπης. Άρα να μην έχουμε μόνο τη φύση στο μυαλό μας. Καλές είναι αρκούδες και ηλίκοι, αλλά να σκεφτόμαστε και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ευχαριστώ κύριε Ντόρφμαν για 1,5 λεπτό. Τζουφρίντα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, καταρχά θα ήθελα να υποφεληθώ από την παρουσία σα να σε ευχαριστήσω για την ευαισθησία και την ετοιμότητα που δείχνετε με τις δηλώσεις σας ε, μετά τον σεισμό στην Κεντρική Ιταλία. Δείξατε ότι είναι διαθέσιμη η Κομισιόν να ετοιμάσει παρεμβάσει ανάλογα με τι ανάγκε των περιοχών αυτών που επλήγησαν και υπέστησαν τρομερές ζημιές και σε ζωές και σε κτίρια. Θα πρέπει να υπάρχει η πολιτική αυτή, ε, η πολιτική αυτή να, είναι, να δημιουργήσει απασχόληση, αλλά θα πρέπει να είναι στατική. Δεν θα πρέπει μόνο να βασιστούμε στον βιομηχανικό ιστό. Ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η βάση αυτού του ιστού, κυρίως ε, σε Περιοχέ όπου δεν υπάρχει τέτοια μεγάλη ανάπτυξη όπω ο τη Ιταλία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσει είναι ε, η ατμομηχανή τη οικονομία μα. και προ εκεί λοιπόν θα πρέπει να στραφεί η πολιτική συνοχή. Αλλά συχνά η πραγματικότητα μα λέει ότι τα αντιδραστικά ταμεία δυστυχώς ε, δεν είναι για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, γιατί υπάρχουν τεράστιοι φραγμοί να υπερβληθούν, κυρίω τη γραφειοκρατία και την πρόσβαση στην πίστοση. Όπως ε, πολύ σωστά είπε η έκθεση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίσουν πάρα πολλά φράγματα λόγω της περιπλοκότητας του συστήματος προγραμματισμού σε όλες τις φάσεις. Επίσης, η πρόσβαση στην ε, πίστη είναι πολύ σημαντική για την, ε, ε και για την πολιτική συνοχή, ε, αλλά και τα νέα χρηματοδοτικά μέτρα θα, θα δώσουν τη δυνατότητα και στις τράπεζες να απελευθερώσουν νέα κονδύλια. Χάρη σε αυτά τα λεφτά θα μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν ανάπτυξη και να παράγουν πλούτο. Ευχαριστώ, Τζούλι Γκόρτ, για 1,5 λεπτό. Um, first of all... Πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο ε, σχετικά ε, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η σπονδυλική στήλη ε, της οικονομίας μας. Θα μπορούν ε, να εμπορεύονται, να εργάζονται σε όλη την Ευρώπη, κυρίως στο δημιουργικό τομέα, στον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Κάθε στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει εναλλακτικά μοντέλα επιχειρήσεων, διότι έχουν τόσες πολλές δυνατότητες ε, για επιχειρηματικότητα και μπορούν να φέρουν ανταγωνιστικότητα στον ιδιωτικό τομέα. Ε, θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση, στην επιχειρηματικότητα, κυρίως οι γυναίκες και τα κορίτσια, τα οποία έχουν αντιμετωπίσουν προκαταλήψεις. Η ανάγκη καινοτομία και ε, συνέργειας με την στρατηγική της κοινοτομίας είναι σημαντική. Ε, πρόκειται για μια εγκάρσια αντίληψη η καινοτομία. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των μέσων χρηματοδότησης που είναι ε, κρίσιμα κυρίως ε, στην Ήπεθρο. Πέρσι τον Ιούλιο συμμετείχα στο φόρουμ στο Μάντσεστερ για την επιστήμη στην εκλογική μου περιφέρεια όπου είδαμε τι μπορεί να προσφέρει η επιστήμη με τη συνάδελφα Βεν και θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Οι επιχειρήσεις, οι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες όλοι ήσαν υπέρ μιας πιο συνολικής προσέγγισης στην καινοτομία και στην αποκοινού διερεύνηση της επίπτωσης πάνω στην κοινωνία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, υπέρ ειδίκευσης, εξειδίκευσης. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Τσάμπα Μόλντα. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πολιτική συνοχή και σε όλα αυτά τα προγράμματα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι η διαφθορά. Υπάρχει μια σειρά κρατών μελών ε, όπου έχουμε, ακούμε πολλά για τη διαφθορά. Το χειρότερο παράδειγμα είναι η Ουγγαρία, η χώρα μου. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει μία μέρα που να περνάει χωρίς ο τύπος να αναφέρει ένα θέμα που σχετίζεται με έναν πολιτικό, με έναν ολιγάρχη, με ε, μια υπόθεση ε, διαφθοράς. Οι περιπτώσεις αυτές διαφθοράς δεν παρακολουθούνται, δεν διώκονται και δεν υπάρχουν ε, πίνες και κυρώσεις. Υπάρχουν λοιπόν κράτη-μέλη όπου ε, οι εισαγγελείς φαίνονται να ασχολούνται με τα θέματα της διαφθοράς, αλλά δεν κάνουν και πολλά πράγματα. Τα κράτη-μέλη τα οποία πραγματικά αντιτίθενται στην ε, δημιουργία μιας εισαγγελία για την Ευρώπη είναι αυτές οι οποίες φοβούνται ότι θα μπορούσε αυτός ο θεσμός να παρέμβει στις δικές τους υποθέσεις. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Αν μια κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει για να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό γραφείο εισαγγελέως, τι σημαίνει αυτό. Διότι δεν θέλουν αυτές οι περιπτώσεις διαφθοράς να διώκονται, να ερευνώνται. Εξού και η σύστασή μας, ίσως όχι τώρα, αλλά μετά το 2020 και την περίοδο συνοχής μετά το 2020 θα πρέπει να πούμε ότι μόνο τα κράτη-μέλη που είναι έτοιμα να υποστηρίξουν την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα υποστηρίζονται, θα βοηθούνται. Όλοι θέλουν να πάρουν τα χρήματα, αλλά δεν θέλουν να διώκονται αυτές οι περιπτώσεις. Ευχαριστώ Κατζιάη. Έχω διπλάσιες αιτήσει από χρόνο, οπότε θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που δεν έχουν μιλήσει ακόμα στη διαδικασία Catch και που ήταν παρόντες καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Ο κύριος Νόβακοφ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το να έχεις γεννηθεί στα Βαλκάνια δεν είναι πάντα δυστυχία. Γιατί η δύσκολη πραγματικότητα σε κάνει ευφυή, δημιουργικό, ευρηματικό για να αντιμετωπίσεις τα δύσκολα προβλήματα. Άκουσα φωνές εδώ ε, που μιλάνε για τον περιορισμό της πολιτικής συνοχής. Κοιτάξτε, η πολιτική συνοχή δεν είναι ένα κέικ που το κόβουμε κομματάκια όπως θέλουμε. Υποστηρίζεται και από τους εθνικούς προπολογισμού και από τις εθνικές πολιτικές και υπάρχουν εκατοντάδες περιφέρειες που βασίζονται σε εμά. Τι θέλουμε, θέλουμε να αυτοπυροβοληθούμε. Επομένως, αυτά τα άτομα τα οποία λένε να περιορίσουμε την πολιτική, τι θα γίνει αν το κάνουμε αυτό κύριε και κύριοι. Νομίζω ότι είναι κενά λόγια. Αρκετά ακούσαμε τέτοιου τύπου λόγια. Βέβαια έχουμε ακούσει τα πάντα εδώ μέσα. Αλλά ελπίζω η φωνή των περιφερειών να πριτανεύσουν. Οι φωνές των περιφερειών να πριτανεύσουν πολλοί έχουν το βλέμμα στραμμένο πάνω μας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, γραφειοκρατία και ελπίζω να πρετανεύσει λογική τελικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νοβακόφ. Η κυρία Γκραπίνη, παρακαλώ. Domnule președinte, doamna comisar, uh, apreciez foarte mult dezbaterea de astăzi pentru Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, εκτιμώ πολύ τη συζήτηση που κάνουμε απόψε διότι θεωρώ ότι για την Ενωμένη Ευρώπη η συνοχή έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό. Θέλω να αναφερθώ λίγο στην έκθεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί είμαι και πρόεδρος ε, σε μια διακομματική ομάδα, ένα intergroup για τις μικρομεσαίες. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέμε, κύρια Επίτροπε, ε, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε γιατί οι μικρομεσαίες ε, επενδύσεις δεν έχουν πρόσβαση ε, στις δημόσιες επιχειρήσεις, σε δανειοδότηση, στην έρευνα και την καινοτομία. Όταν μιλούμε για συνοχή θα πρέπει να ξέρουμε και τι γίνεται με το σχέδιο στρατηγικών επενδύσεων που δεν χρησιμοποιείται για τη συνοχή. Και αυτό οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες που εντείνονται μεταξύ των περιφερειών. Γι' αυτό κυρία Επίτροπε σας παρακαλώ πάρα πολύ να φροντίσετε ε, έτσι ώστε μέσω πρόθεσμα να αντιμετωπιστεί και αυτό το θέμα, μήπως χρειάζεται να γίνουν και κάποιες αλλαγές. Και βεβαίως προφανώς θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τις ναυφείς επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας στις παραμεθόριες περιοχές και όχι μόνο. Και διασυνοριακά υπάρχει συνεργασία ε, ακούγονται διάφορα προγράμματα και έργα, το είπαν και συνάδελφοι. Γι' αυτό ελπίζω να συνεχιστεί η συνοχή και να είναι ε, θεμέλιος Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, η καινοτομία δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο ότι μια αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να αλλάξει τον τρόπο διακυβέρνησής της. Οι περιφέρειες, οι ε, περιοχές που αναπτύσσονται έξυπνα ε, προωθούν την καινοτομία και καθώς αδυναμώνονται και καθώς δημιουργούνται φυσικές συνέργειες αποδεικνύεται ότι η προστατευτική κρατική λογική δεν είναι καλύτερη για να προωθήσει μια παραγωγική οικονομία. Χαίρομαι που η Κομισιόν Ενστερνίζεται ε, αυτή τη λογική όλο και περισσότερο για τις ευρωπαϊκές ε, περιφέρειες, ούτως ώστε να υπάρξουν στρατηγικές ε, έξυπνης εξειδίκευσης. Δεν θα πρέπει να χάσουμε το τρένο τη ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε αυτή την ικανότητα στρατηγική δράση. Να βελτιώσουμε τη θέση μα. Αυτή είναι η βάση για τη δημιουργία και ποιοτικών θέσεων απασχόληση. Αυτέ θα πρέπει να είναι οι πολιτικέ μα και οι διεκδικήσει μα και αυτέ είναι ούτω ή άλλω ω χώρα. Εμεί ω Ισπανία αυτά ζητάμε. Ευχαριστώ κύριε Πελπάου. Ο συνάδελφο Βίγκα. Senhor Presidente, falo num período onde prossegue uma uma inaceita, inaceitável chantagem da Comissão. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε σε μια φάση απαράδεκτου εκβιασμού απέναντι στη χώρα, στη μας από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκβιάζει την Πορτογαλία. Το 2015 εκλέξαμε μία κυβέρνηση, νόμιμη κυβέρνηση, αλλά σταμάτησε η δράση της λόγω των ε, εκβιαστικών πολιτικών της Τρόικας συνεχίζεται αυτός ο εκβιασμός. Τώρα οι Βρυξέλλες δείχνουν το πραγματικό του ε, πρόσωπο. Ε, και πώς θα διορθώσουν τις ε, εθνικές και περιφερειακές ασυμμετρίες. Αντί να αναγνωρίσουν ότι ατύχησαν αυτές οι πολιτικές, η Κομισιόν προσπαθεί να τιμωρήσει τώρα την Πορτογαλία και άλλες χώρες, ακόμα περισσότερο, τις χώρες μάλιστα που επλήγησαν πολύ περισσότερο από τη λιτότητα. Και με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ορθοποδήσει η οικονομία μας. Ευχαριστώ. Συνάδελφος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν τον σημαντικότερο κινητήρα ανάπτυξης διότι έχουμε 100 εκατομμύρια άτομα και 85% των νέων θέσεων εργασίας. Στην Γαλλία είναι 3,5 εκατομμύρια μικρομεσές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δίνουν δουλειά σε 6 στα 10 άτομα. Ήμουν επικεφαλή μια μικρή επιχειρήση και διαπίστωσα ότι πολύ συχνά οι προτάσει πολιτικέ είναι μακριά από την πραγματικότητα των επιχειρηματιών. Βεβαίω η έκθεση αυτή κάνει καλέ διαπιστώσει και καλές προτάσεις, αλλά ας ξεχάσουμε τις ε, ιδεολογικές ε, διαφορές. Ε, ας επιδείξουμε ρεαλισμό και καινοτομία ούτω ώστε το πολιτικό στοιχείο να μην καθυστερεί σε σχέση με το οικονομικό. Οι πολιτικοί δεν θέλουν μόνο να επιβάλλουν νόμους, φόρους, να δίνουν ε, επιδοτήσεις, ε, θέλουν οι μικρομεσαίες σταθερό φορολογικό περιβάλλον, λιγότερο διοικητικό φόρτο, καλύτερη πρόσβαση στις πιστώσεις ε, και απέναντι στο dumping καλύτερη προσέγγιση. Ευχαριστώ. Αυτές είναι οι προτάσεις. Ευχαριστώ κυρία Μπίλντε. Τελευταίος ο κύριος Συναδεινός. Κύριε Πρόεδρε, η της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι αποκλειστικά θέμα χρηματοδότησης όσα χρήματα και αν επενδυθούν δεν θα φέρουν από μόνα του την ανάπτυξη. αν ήταν τόσο απλό τα δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν αποδοθεί από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία θα έπρεπε να μεταφράζονται σε μειωμένου δείκτε ανεργία και εσωτερική μετανάστευση. η ένωση πρέπει να υιοθετήσει μέτρα και κανόνε που ευνοούν τη σύσταση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στηρίζουν την επιβίωση αυτών εντό του ανταγωνιστικού περιβάλλοντο με τι μεγάλε επιχειρήσει. θα αναφερθώ σε τρία απλά μέτρα κατάργηση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων σύσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θεσμοθετώντα ένα πανευρωπαϊκό πρότυπο μια οδηγία εφαρμόσιμη από όλα τα κράτη μέλη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντο προ δύο κατευθύνσει μετάβαση προ μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και προώθηση πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών συνδυασμό των διορθωτικών ταμείων με άλλου πόρου που θα ευνοήσουν τον τραπεζικό δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. τέλο ανάπτυξη μιας ενιαίας φορολογικής πρακτικής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα επιτρέπει τη φορολόγηση μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο χάριτος ή θα επιβάλλει ενιαίες φορολογικές κλίμακες από όλα τα κράτη μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Συνέδρινε. Ολοκληρώνεται εδώ η διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ και για να κλείσει η κοινή συζήτηση θα λάβει το λόγο ξανά τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά οι εισηγητές. Η κυρία Κρέτσου πρώτη, κυρία Επίτροπος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης ιδιαίτερος τους ε, βουλευτές για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πολύ χρήσιμα όσα μας είπατε και τα όσα ακούσαμε εξ ονόματος των επιμέρους επιτροπών ε, ε, του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάρα πολλοί ομιλητές αναφερθήκατε σε αυτές. Και πραγματικά η πολιτική συνοχή θα πρέπει να είναι πάντα προς το συμφέρον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διότι Αυτές είναι πραγματικά η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ως γενική παρατήρηση θα ήθελα να πω εισαγωγικά ότι χάρηκα πάρα πολύ ε, που οι περισσότεροι ομιλητές ετώνησαν την πολιτική της συνοχής. Παρά ε, ορισμένες επικρίσεις που ακούστηκαν για ε, ορισμένες ελλείψεις και κενά που πρέπει να καλυφθούν. Είναι γεγονός αυτό, αλλά η πολιτική συνοχής θα πρέπει να σημαίνει ουσιαστικά βελτίωση της καθημερινότητας κάθε πολίτη. Και είναι πολύ σημαντική για όλα τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Για τις μικρομεσαίες έχουν διατεθεί μέχρι το 2020 90 δισεκατομμύρια ευρώ και ελπίζω να αντλήσουν τα κονδύλια αυτά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι εμείς κάναμε πολλές προσπάθειες ουσιαστικές για να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και το φόρτο για τις επιχειρήσεις. Τα προγράμματα να ε, απορροφώνται και να εκτελούνται καλύτερα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα στο μέλλον και να συνεργαζόμαστε με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές σας. Ως γνωστό έχετε την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιτροπή για ε, τον έλεγχο των προπολογισμών και οι επιτροπές αυτές καλύτερα μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση του κυρίου Βαλκάρθελ, βεβαίως ε, θέλουμε να πετύχει πολιτική συνοχής και σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά για την έρευνα και την κοινοτομία και την έξυπνη εξειδίκευση. Όσοι ενδιαφέρονται άμεσα ε, δεν είναι μόνο οι πρόσωποι της τοπικής και περιφερικής ε, αυτοδιοίκησης αλλά και εκπρόσωποι πανεπιστημίων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνεργάζονται για την έξυπνη εξειδίκευση. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύνδεσμο για τη συνεργασία αυτή, μια δικτύωση ουσιαστικά για την καλύτερη χρήση και των ενεργειακών πόρων, αλλά και αλλού στα τρόφιμα, ε, στη μηχανική. Ε, μπορεί να βοηθήσει μια τέτοια δικτύωση και μια συνεργασία. Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί κάθε περιφέρεια να γίνει Silicon Valley. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλουμε είναι να αναπτύσσονται ακόμα και οι πιο καθυστερημένες περιφέρειες τα χρήματα ε, που διατίθεται μπορούν να πιάσουν τόπο. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρωτοβουλία της κυρίας Μιχαήλοβα για την εδαφική συνεργασία, καλωσορίζω ε, τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά και υπάρχει το πρόγραμμα Interreg το οποίο μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα προς μίμηση για να αποδείξουμε τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Το 25% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε παραμεθόριες περιοχές. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διασυνοριακή συνεργασία πασθησία. Υπάρχει ήδη πολύ καλή συνεργασία, ε, για παράδειγμα, μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας αλλά αντίστοιχα θα μπορούσαν η Γαλλία με το Βέλγιο να συνεργάζονται καλύτερα. Τη στιγμή που η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο. Για να γίνει αυτό πρέπει να ε, εφαρμόζεται μια νέα νομοθεσία προσαρμοσμένη ε, να αποδομούνται τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ιδιαίτερα σε καιρούς δύσκολους που έχουν επανέλθει οι έλεγχοι στα σύνορα. και ε, μπορεί, η πολιτική με τη δράση της να βοηθήσει την ανάπτυξη των περιφερειών. Σας μίλησα για το Interreg. Έχουμε την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και βρισκόμαστε ήδη στο πέμπτο πρόγραμμα Interreg. Ε, εργαζόμαστε αυτό το καιρό για να προετοιμάσουμε τα επόμενα προγράμματα, το έκτο Interreg. Έρχομαι τώρα στην έκθεση της κυρίας Μπρέσο για τη στρατηγική των Άλπαιων. Και η κυρία Μπρέσο τόνισε προηγουμένως ότι η στρατηγική για τις Άλπες ε, ε, θα πρέπει να είναι σημαντικό στοιχείο για την ε, εδαφική συνεργασία. Τους επόμενους μήνες θα δημοσιεύσουμε μία έκθεση εξαμήνου για την μακροπεριφερειακή στρατηγική όπως ε, ζητεί και ίδια στην έκθεσή της και θα αξιολογούμε εκεί την ευρωπαϊκή στρατηγική και για την περιοχή των Άλπαιων και για τον τρόπο με τον οποίο στο μέλλον θα πρέπει να διαμορφωθεί η εδαφική συνεργασία έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να δουν να βελτιώνεται το ιδιωτικό τους επίπεδο ακόμα και στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες. Στην παρούσα φάση λοιπόν δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις γιατί έχω και περιορισμένο χρόνο αγόρευσης. Είναι και τέσσερις εκθέσεις. Δεν μπορώ να καλύψω όλα τα θέματα. Και για να μην αδικήσω κανέναν ε, θέλω να πω ότι μίλησε ο κύριος Φουντούλης ε, από την Ελλάδα. Μια χώρα που έχει πάρει τόσα εκατομμύρια και λέγει ότι η πολιτική συνοχής αφορά μόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ε, σας προτείνω να πάμε μαζί στην Ελλάδα για να δούμε πόσο χρησιμεύει η πολιτική συνοχής και τι ωφέλεια υπήρχε για την Ελλάδα. Έκτακτα μέτρα που λάβαμε σε έκτακτες περιστάσεις και καμία άλλη χώρα δεν έχει λάβει τόσα κονδύλια από την πολιτική συνοχή όσο η Ελλάδα. Και... αν δεν έδινε τη χρηματοδότηση κατά 90% η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε η Αθήνα ε, να κάνει αυτά τα έργα. Και στην Θεσσαλονίκη είχαμε χρηματοδότηση ευρωπαϊκή για τα σχολεία ε, που αποκαταστάθηκαν. Θυμάστε ποια ήταν η Ελλάδα, τι εικόνα είχε πριν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βελτίωσε σημαντικά τη θέση της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των ετών. Συνεισέφερε σημαντικά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουμε εργαστεί προς το συμφέρον της Ελλάδας. Και τελικά είναι άδικη αυτή η κριτική την οποία μας απευθύνεται. Κάναμε πολύ σημαντικά πράγματα για να βελτιωθεί η ζωή των Ελλήνων πολιτών. Ήθελα να το πω αυτό στο τέλος να το τονίσω. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Μαδέρα και την Ιταλία, ε, για τα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι, τις θεομηνίες αυτές, θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς ε, τους κατοίκους των περιεχών αυτών. Μέσα Νοεμβρίου θα έχουμε τη δυνατότητα να κινητοποιήσουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης. Πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ ε, έχουν ε, προβλεφθεί για την Ιταλία για την πρόληψη των θεομηνιών. Και το 2009 ήδη, μετά το σεισμό στο ε, Άκουιλα, ενώ το 2012 ε, είχαμε κι άλλο σεισμό στην περιφέρεια Εμίλια Ρωμάνια. Τι έγινε με όλα αυτά τα προγράμματα για την πρόληψη των θεομενιών και στην Ιταλία. Αν χρειαστεί μπορούμε να τερματίσουμε, να αλλάξουμε μάλλον το ΕΣΠΑ για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ιταλία, αλλά Υπάρχουν ήδη πολλά χρήματα που διατίθεται για την Ιταλία για την πρόληψη αυτών των καταστροφών. Ξέρουμε ότι η οροσυρά των Απενίνων δυστυχώς είναι σεισμογενής. Οπότε, στην ετήσια σύνοδο των περιφερειακών ε, των απομακρυσμένων περιφερειών θα το συζητήσουμε και αυτό ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη στήριξη της μαδέρας. Αλλά θα πρέπει τις αποφάσεις να τις παίρνουμε από κοινού με τις ε, τοπικές αρχές. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικές, με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κατάγονται από τις περιφέρειες αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αναφερθήκατε στον συνάδελφο Φουντούλη, ο οποίο δυστυχώ έχει αποχωρήσει. Καμία φορά καλό θα ήταν οι συνάδελφοι που μολούν και αποχωρούν να μην δέχονται και ιδιαίτερη τιμή να αναφερόμαστε σε αυτό στη συνέχεια. Ε, υπο, ε, τώρα, για δύο λεπτά η κυρία Νταμάτο πρώτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μετά από τη συζήτηση θα ήθελα να ξανασταθώ σε κάποια βασικά για μένα θέματα. Η οικονομική κρίση έγινε αλλά κυρίως η πολιτική λιτότητα ε, στράγγλισε την εσωτερική ζήτηση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να τις βοηθήσουμε και να τους δώσουμε πρόσβαση στην ε, πίστοση. Θα πρέπει να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε τη σχέση ανάμεσα στο τραπεζικό σύστημα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το χρηματοδοτικό σύστημα ε, είναι τέτοιο που δεν βοηθούν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη, στο χρήμα και στις επιδοτήσεις. Ε, εμείς δεν συμφωνούμε με την αισιοδοξία της Κομισιόν για την ε, ένωση των κεφαλαίων αγορών. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη διαφάνεια στην χρήση των πόρων. Να συμμετάσχουν ακόμα περισσότερο οι τοπικές αρχές, οι επιχειρηματίες, στο, στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων ούτως ώστε να προωθήσουμε κάποια έργα, ούτως ώστε να λάβουμε ε, υπόψη τις ανάγκες των τελικών δικαιούχων. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την αρχή της εταιρικής σχέσης και να αποφύγουμε ότι η πολιτική συνοχή θεωρείται ως μια επιπλέον επιβολή εκ των άνω. Είναι πάρα, πολύ, πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να βελτιώσουμε. Ε, έχει μεγάλη ευθύνη εδώ το κάθε κρατός μέλος, κυρίως της Νότιας Ευρώπης, που ε, εποφελήθηκαν μέχρι στιγμής από την πολιτική συνοχή. Πολλά όμως από αυτά τα κράτη δεν έχουν ε, εκφράσει ξεκάθαρη θέση ακόμα. Ε, το βασικό είναι όμως το Horizon 2020 ε, να προωθήσει πιο απλά έργα και δεν καταλαβαίνουμε γιατί μερικές φορές θεωρούνται κακά αυτά τα έργα τα οποία προωθούνται από τον ορίζον 2020. Η πολιτική συνοχή είναι το μόνο πραγματικά δημοκρατικό εργαλείο και προωθεί μια ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κ. Βαλκάσελ Σίσο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι για τη θετική αξιολόγηση που έκανε η Κομισιόν για την ε, δική μου έκθεση, για το ΡΙΣΤΡΙΑ. 3. Χαίρομαι επίσης για αυτό που είπατε για τους ε, οδηγούς καλών πρακτικών, για την ε, διαμόρφωση και την ανάπτυξη αυτών των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης και για τις προσπάθειες που κάνετε από πλευρά Επιτροπής για να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και μεταξύ των προγραμμάτων διεθνικής συνεργασίας, ούτως ώστε να βελτιστοποιήσουμε τους πόρους και να αποφύγουμε τις αλληλεπικαλύψεις. Τέλος, η συνοχή φτιάχνει αυτοκινητοδρόμους, σηκώνει ε, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά κέντρα, σχολεία κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και τα χρειαζόμαστε. Και οι η Ισπανία υποφελήθηκε από αυτές τις ε, πολιτικές. Αλλά το βασικό είναι να έχουμε και αυτοκινητόδρομου ε, που να συνδέουν τους λαού μα. Και τι είναι αυτό που απομακρύνει τους λαού, είναι η έλλειψη γνώση. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν τεχνολογική ε, ανάπτυξη, έρευνα, δηλαδή αυτή είναι η βάση που υποστηρίζει αυτές τις στρατηγικές ε, ανάπτυξη. Και η γνώση είναι ο αυτοκινητόδρομο του μέλλον. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βάλκαρ Σελσίσο. Η κυρία Μιχαήλοβα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας σχετικά ε, με την ε, δική μου έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εξέφρασαν τις απόψεις τους ε, στην Επιτροπή Ρέτζη Εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά για αυτήν την έκθεση. Θα ήθελα να τονίσω άλλη μια φορά ότι έχει αποδείξει η πολιτική αυτή τις δυνατότητες και την δύναμή της, όχι μόνο για τα εδαφικά, αλλά και σε τομείς ως η ψηφιακή τεχνολογία, ενέργεια, η επιστημονική έρευνα, η, η έξυπνη εξειδίκευση στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος κλπ. κλπ. Είμαι, ε, νομίζω ότι μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η πολιτική αυτή στην πολιτική συνοχή μετά το 2020 νομίζω ότι η εδαφική πολιτική μπορεί να γίνει η βάση για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δυνατότητες των διαφόρων περιφερειών και εδαφών ανεξάρτητα για το τι μιλάμε, αν μιλάμε για διασυνοριακές περιοχές ή άλλα εδάφη, η εδαφική συνεργασία έχει μεγάλη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και είμαι πεπισμένη ότι τέτοιες συζητήσεις όπως αυτή που είχαμε σήμερα θα αναπτύξει την ολοκληρωμένη εδαφική συνεργασία. Ευχαριστώ κυρία Μιχαέλοβα. Και τώρα δίνω τον λόγο στον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο, την κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους, ευχαριστώ και την Επίτροπο για τις ενδιαφέρουσες αναγγελίες που μας έκανε για το μέλλον των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και κυρίως της δικής μας περιφέρειας. Για τη δική μας περιφέρεια. Η πρόκληση θα είναι, το είπα και προηγουμένως, να κρατήσουμε ενωμένη αυτή την πολύ διαφορετική περιφέρεια. Υπάρχουν κάποια σημεία της περιφέρειας που είναι πολύ ανεπτυγμένα, κάποια που αντιμετωπίζουν μεγάλη μόλυση, άλλα σημεία που έχουν οικονομικές δυσκολίες δεν θα πρέπει να εμπλέκουμε μόνο τις ε, πρωτεύουσες, αλλά και τις απομακρυσμένες περιοχές, τα, και την Παιδιάδα και τις, τα βουνά. Η πεδιάδα ε, πάντα έχει αυτή τη δυνατότητα καινοτομία. Και επίση στις ορεινές περιοχέ θα πρέπει να του βοηθήσουμε να φτιάξουν και να προωθήσουν νέα έργα, ούτω ώστε να μην υπάρχουν πολίτε κατηγορία Α και κατηγορία Β. Εδώ μπορούν να μα βοηθήσουν οι νέε τεχνολογίε με τηλεργασία ας πούμε. Υπάρχουν νέες ε, ευκαιρίες εργασίας. Θα ήταν πολύ καλό αυτό για την περιοχή των Άλπαιων. Επίσης η εκπαίδευση εξ αποστάσεως, πολύ ενδιαφέρουσα. Όλα αυτά θα βοηθούσαν ε, μια τόσα δύσκολη και περίπλοκη περιοχή όπως αυτή των Άλπαιων. Ακούστηκαν διάφορες παρεμβάσεις για το Τωρίνο Λιόν, για τη γραμμή αυτή τη ισοδομική. Η γραμμή αυτή δεν αφορά, δεν συζητάται σε, μία, σε αυτή την γνωμοδότηση, σε αυτή την έκθεση. Έχει αποφασιστεί και υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Εμεί μιλάμε στη δική μα γνωμοδότηση για την ανάγκη αυτά τα μεγάλα έργα να εξασφαλίσουν τι διασυνδέσεις σε όλη την αλπική και περιαλπική περιοχή, ούτω ώστε να αξιοποιήσουμε την περιοχή αυτή, την περιφέρεια αυτή. Και τέλος πάντων αυτή είναι μια ουσιαστική γραμμή για να μειώσει την κυκλοφορία με τα αυτοκίνητα και την κυκλοφορία των φορτηγών. Και επίσης και στον Κοτάρντο ε, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε ότι η μεγάλη κίνηση των αυτοκινήτων γίνεται μέσω του Κοτάρντο. Ευχαριστώ κυρία Μπρεσό. Ολοκληρώνεται εδώ κοινή συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι έκθεση του κ. Κοράου και αφορά το καταπιστευματικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική, επιπτώσει για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Το λόγο έχει πρώτος ο εισηγητή, ο κύριος Κοράου, για τέσσερα λεπτά παρακαλώ.